Good afternoon, dear colleagues, dear guests. Αγαπητοί φιλοξενούμενοι, αν θέλετε καθίστε. Για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Έγκριση της σας διάταξης, πρώτο θέμα. Σας παρακαλώ καθίστε. Uh, λοιπόν, όσον αφορά την ημερήσια διάταξη, το σημείο 3 που είναι η έγκριση των πρακτικών, το 7, την κοινή ομάδα επιχειρησιακή ΜΑΡΕ, μετά συμφωνία ΕΠΑ Ευρωπαϊκής Ενώσεως για προστασία προσωπικών δεδομένων από το επόμενο σημείο, σημείο 9, Λοιπόν, ε, προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά πρέπει να αναβληθούν τα σημεία αν δεν έχετε αντίρρηση, εγκρίνεται τροποποιημένη η ημερήσια διάταξη. Τώρα, για τη διερμηνία. Δανέζικα, λετονικά, κροατικά, δυστυχώς δεν έχουμε. Και έχω μακρά λίστα για την έγκριση συστάσεων των συντονιστών. Πρέπει να διαβάσω όλες τις αποφάσεις των συντονιστών. Για το διορισμό εισηγητού για γνωμοδότησης, η κυρία Γκέμπριελ του ΕΛΚ διορίστηκε εισηγήτρια όσον αφορά την σύναψη συμφωνιών από θεώρηση μεταξύ αντολικό Τιμόρου, Αντομινική Δημοκρατία, Σεν Βίνσεν Γρεναδίνε, Σαμόα, τον Μπάγκο, την Ιδάδ Βανουά του Γρενάδα, προσωρινή άρση τη απέτσια θεώρηση. Δεύτερη πρόταση γνωμοδότηση, πρόταση για οδηγία του Συμβουλίου, τροποποιεί την οδηγία που αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των φορολογικών. Εδώ οι συντονιστέ αποφάσισαν ότι καμία γνωμοδότηση δεν πρόκειται να συνταχθεί. Όμω τροπολογίε μπορούν να υποβληθούν άμεσα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Μετά, όσον αφορά τι ακροάσει και αποστολέ για το δεύτερο εξάμεινο του 2015, οι συντονιστές ενέκριναν τον κατάλογο των ακροάσεων και των αποστολών για το δεύτερο εξάμεινο και αυτός ο κατάλογος διενεμήθη προς τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, Ευρωπαϊκός σε αιτήματα για συμπερίληψη του δημοσίου καταλόγου των πρακτικών συνεδριάσεων συντονιστών των επιτροπών για την περίοδο 2009-2014 οι συντονιστές συμφώνησαν, υπάρχει πρόταση από τα στοιχεία, στη δημοσίευση όλων των υφιστάμενων σημειώσεων που υπήρχαν ε, και υπάρχουν στο αρχείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καθορισμός παρατηρητού για την εκλογή του Προέδρου του Eurojust 21 Απριλίου του 2015. Οι συντονιστές αποφάσισαν να στείλουν ένα μέλος της γραμματείας της ΛΥΜΠΕ που θα είναι παρατηρητής, ε, κάτι το οποίο έγινε και κατά το παρελθόν. Μετά έχουμε σχέδιο επιστολής Προέδρου προς την Προεδρία όσον αφορά τον κανονισμό για νέες ψυχότροπες ουσίες και την οδηγία που τροποποιεί την, απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου που αναφέρει τα βασικά συστατικά των ποινικών πράξεων και των αδικημάτων όσον αφορά το παράνομο εμπόριο των ναρκωτικών. Οι συντονιστές συμφώνησαν να αποσταλεί αυτή η επιστολή στην Προεδρία του Συμβουλίου οι συντονιστέ συμφώνησαν να διοργανωθεί δομημένο διάλογο όπω προβλέπεται στα πλαίσια τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη συνάντηση με τον Επίτροπο Αβρομόπουλο και Ζούρβα με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαν θα μπορούσε να λάβει χώρα 6 και 7 Μαΐου του 2015. Μετά έχουμε την κοινή επιχειρησιακή ομάδα ΜΑΡΕ που ζητήθηκε να προσθεθεί στο πρόγραμμα της ΛΥΜΠΕ του Απριλίου σαν σημείο ενημέρωση από πλευρά Ευρωπόλ και Επιτροπής, οι συντονιστέ συντονιστές αποφάσισαν το θέμα αυτό να τεθεί στην ημερήσια διάταξη της ε, ΛΥΜΠΕ και μετά οι συντονιστέ συνέστησαν τι τις κάτωθι προτάσεις ψηφίσματος που δεν θα πρέπει να βρουν συνέχεια. Γιακοβιτ, το Ευρωπαϊκό Έτο του Παιδιού, χάρη, ε, μπιζότο για την αύξηση των περιπτώσεων ε, φοβισμού στο διαδίκτυο στην Ιταλία, Μπιζότο για την δίσδυση των τρομοκρατών στην Ιταλία μέσω παράνομη μετανάστευση και Μπιζότο για την ε, τα νέα συνθετικά ναρκωτικά που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, μπιζότο παράνομο εμπόριο ανθρώπινων οργάνων από την Αφρική και ξανά μπιζότο για τη διαμαρτυρία μεταναστών στο Βιτόριο Βένετο. Μετά δύο προτάσεις Γιάκοψη, τις προτάσεις για τη βία στις αθλητικές εκδηλώσεις και για την διάλυση των διαφόρων ιδρυμάτων για τη αιμονή παιδιών. Μετά έχουμε τις αναφορές να μην συνεχιστούν που πρότειναν συντονιστέ. Αναφορά της κυρίας Ουγγάρος, αναφορά τον εκλογικό νόμο στην Ουγγαρία, Σάρα Λουζία Χάσελ Ρόιζινγκ όσον αφορά την τροποποίηση της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και επίσης ε, μια άλλη αναφορά που υπευλήθη από τον κύριο Φλάβιο Μικόν όσον αφορά τη δικαιοσύνη στην ε, Ιταλία. Σας διάβασα λοιπόν ε, όλες τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές. Το ερώτημά μου είναι κατά πόσο η Επιτροπή συμφωνεί με τις προτάσεις αυτές των συντονιστών. Μάλιστα συμφωνείτε και σας ευχαριστώ. Και τώρα πάμε στο σημείο τέσσερα αμέσως πάμε στη συζήτηση όσον αφορά τις, τους όρους για είσοδο και διαμονή υπηκών τρίτων χωρών για λόγους έρευνας, μελετών, σπουδών, ανταλλαγής σπιτιτών αμοιβόμενη και μια αμοιβόμενη κατάρτιση, εθελοντική υπηρεσία όσον αφορά τους ΟΠΕΡ. Η κυρία Βίκστρομ είναι η συγγήτρια. Θα ζητήσουμε από την κυρία Βίκστρομ ε, να παρουσιάσει την όλη κατάσταση μετά το δεύτερο τριγωνικό διάλογο που έλαβε χώρα στις 31 Μαρτίου. Έχετε λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ήδη θα αναφέρατε, ε, δεύτερος τριγωνικός διάλογος έλαβε χώρα στις 31 Μαρτίου και συζητήσαμε βασικά όλο το πεδίο εφαρμογή τη ε, οδηγία που συνέχιστηκε προηγούμενο τριγωνικός διάλογος για τι γενικέ συνθήκε και όρου και συγκεκριμένους όρους για τους φοιτητές και τις οικονομικές δραστηριότητες. Πρόσβαση δηλαδή στην νόμιμη εργασία ε, από τους φοιτητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το πεδίο εφαρμογή, όλα τα θεσμικά όργανα επανεπιβεβαίωσαν τις θέσεις τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι θα υπήρχε προστιθέμενη αξία στη νέα πρόταση αν συμπεριλάμβανε τις επιπλέον κατηγορίες ως υποχρεωτικές και επίσης να ε, βάλει και τις, ε, και τις ΟΠΕΡ και την ε, έμιστη κατάρτιση. Οι ΟΠΕΡ, οι εσωτερικές βοηθοί δηλαδή οι άμυστες δεν καλύπτονται από οποιουσδήποτε κανόνες σήμερα και είναι μια πολύ ευπαθής κατηγορία ατόμων που συχνά τους εκμεταλλεύονται λόγω της ευάλωτης θέσης στην οποία βρίσκονται. Η μαθητευόμενοι επαμοιβοί θα πρέπει να συμπεριληφθούν επίσης. Θα πρέπει κανονικά να ενθαρρύνουμε την πληρωμή της ε, μαθητείας και θα ήταν, κρίμα να βάλουμε την ε, άμυστη αλλά όχι την έμυστη μαθητεία σε αυτή την οδηγία. Και επίσης μας μπερδεύει. Ε, νομίζω ότι ο κανόνας θα πρέπει να είναι η απλού... απλότητα. Το Συμβούλιο επιμένει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για κοινού ε, κανόνες παρά μόνο για δύο κατηγορίες, ε, ερευνητέ και φοιτητέ. Καταφέραμε παρόλα αυτά να, να συμφωνήσουμε για το 6-5 σε ένα δηλαδή σε μια συμβαστική θέση, όταν διευκρινίσαμε ότι αυτό αφορά τις αιτήσει από, από άτομα που είναι νόμιμα παρόντα στην ε, επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση. Φερρυπίν στο Πανεπιστήμιο. Το Συμβούλιο δέχτηκε ξανά την επανεισαγωγή του εκτιμώντας 12 που είχε απαλείψει και που ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τους γιατρούς που κάνουν έρευνα ως ερευνητές και όχι ως φοιτητές. Για τις ειδικέ τώρα συνθήκες των φοιτητών. Το Κοινοβούλιο δέχτηκε την τροποποίηση του Συμβουλίου να βάλει την υποχρεωτική κατάρτιση στην έννοια των σπουδών ε, πλήρους, πλήρους χρόνου. Για τις οικονομικές δραστηριότητες, δηλαδή νόμιμη πρόσβαση στην ε, εργασία, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν υποστηρίζουν την ελάχιστη και μέγιστη, το μέγιστο μάλλον όριο, 20 ώρες τη βδομάδα, ενώ το Συμβούλιο θέλει να επιμείνει στις 10 ώρες, όπως έχουν, που ισχύουν και σήμερα. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι δούλευαν πάντα στα μεγάλα πανεπιστήμια στην, στην Ευρώπη, αλλά στη μαύρη. Στους δύο τριμερείς διαλόγους υπήρξε πρόοδος, αλλά περιορισμένη πρόεδρε. Και λυπάμαι γι' αυτό. Γι' αυτό πρότεινα να αναβάλουμε τον επόμενο τριμερή διάλογο και να ενθαρρύνουμε και τις εργασίες σε τεχνικό επίπεδο στο εσωτερικό του Συμβουλίου, ούτω ώστε να μπορέσει το Συμβούλιο να καταλάβει καλύτερα τα βασικά θέματα. Ούτω ώστε οι διαπραγματεύσεις να μην κολλήσουν σε κάθε ανθιπολεπτομέρεια και να μην σημειωθεί πρόοδο στου ε, τριμμένους διαλόγου. Γιατί αν κάνουμε τριμμένους διαλόγου και δεν υπάρχει πρόοδο, χάνουμε χρόνο. Υποστηρίχθηκε λοιπόν η αναβολή ε, και, από το, και από την Κομισιόν. Δεν έχουμε ακόμα ημερομηνία για την επόμενη συνάντηση. Ε, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη συζητούν τα θέματα που τους απασχολούν, τις κόκκινε γραμμές τους και ο τεχνικός διάλογος και οι τριμερείς διάλογοι θα λάβουν χώρα. Θα ενημερώσω λοιπόν την Επιτροπή για όλες τις εξελίξεις και για όλες τις, τα δύσκολα σημεία. Ελπίζω να σημειωθεί πρόοδος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τονίζω τη σημασία αυτής της οδηγίας. Έχουμε εκθέσεις. Παραδείγματο χάρη, μία έκθεση από τη Γερμανία της προάλλες έλεγε ότι το θέμα των, της ρύθμισης της κατάστασης των ερευνητών είναι σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε κύριε Βίξτρο. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες εξέλιξεις για το θέμα αυτό. Θέλει κανένα συνάδελφος το λόγο? Όχι. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια λοιπόν με το θέμα αυτό. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, στο σημείο 5. Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη, σύσταση 2065 του, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Καλέσαμε τον κύριο Μακναμάρα για να μας μιλήσει για την σύσταση αυτή. Τον κύριο Μάικλ Μακναμάρα που είναι εισηγητής στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κοινοβουλευτική Διάσκευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κύριε Μακναμάρα. Ελάτε παρακαλώ, καθίστε. Για την Επιτροπή μας είναι σημαντική η συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Όπως γνωρίζετε, συναδέλφοι, στο ψήφισμα του για την αξιολόγηση της δικαιοσύνης, το Κοινοβούλιο ζήτησε την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης, και γι' αυτό βρισκόμαστε και σήμερα στα πλαίσια αυτού του διαλόγου εδώ και καλωσορίζουμε τον κύριο Μακναμάρα. Και θα θέλαμε να ακούσουμε για την έκθεση σχετικά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη. Έχει άμεση σχέση και με τη δική μας δουλειά ε, στα θέματα αυτά. Έχετε το λόγο κύριε Μακναμάρα. Um, first of Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ ευγενική σας πρόσκληση να έρθω στην Επιτροπή σας σήμερα. Εκτιμώ ιδιαίτερα την ευκαιρία που μου δίνετε, διότι είμαι και εισηγητής και εκ μέρους της Επιτροπής ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, είναι πολύ ευχάριστο για μένα το να μπορώ να, κάνω, να έχω αυτή τη συνεργασία μαζί σας. Καταρχήν, θέλω να πω ότι το Δεκέμβριο του 2013 η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε μια πολύ επωφελή ε, ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Κίνκα Γκόν, την προηγούμενη πρόεδρο, και μετά την έκθεση του Λουί Μισελ για τα θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012. Ε, σήμερα έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω τη δική μου έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εγκρίθηκε από τη δική μας Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης 27 ε, Ιανουαρίου του 2015 και εγκρίθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή ε, στις 6 Μαρτίου στο Παρίσι. Ξεκίνησε η έκθεση αυτή από μια, από μια συζήτηση που έγινε τον Ιουνίο του 2012, μετά από την οποία το Προεδρείο παρέπεμψε το θέμα αυτό στη δική μα Επιτροπή. Κατά τη συνάντηση αυτή, τα μέλη τη κοινοβουλευτική διάσκεψη ε, εξέφρασαν τι ανησυχίε του για την επικάλυψη που γίνεται στο Συμβούλιο τη Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίως ε, μετά τον διορισμό του ε, ειδικού εκπροσώπου ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακολουθήσαμε στενά τις εξελίξεις για να μπορούμε να παρακολουθούμε το κατά πόσο τηρούνται τα κριτήρια της Κοπενχάγης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Οκτώβριο του 2013 έγινε μια συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να έχουμε συνέργεια και όχι επικάλυψη και εγκρίθηκαν τα, ε, οι συστάσει με βάση την έκθεσή μου. Η συνέλευση επανέλαβε ότι πρέπει να αποφεύγουμε την επικάλυψη εργασιών στο Συμβούλιο της Ευρώπης ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τέτοιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον προϋπάρχοντα ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης που αποτελεί ε, και σημείο αναφορά για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη. Στην έκθεσή μου, εγώ εστιάζω στον τρόπο με τον οποίο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά και, άλλες, και άλλα όργανα, οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πώς λαμβάνουν υπόψη το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης και πώς το προωθούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτά τα στοιχεία, ιδίω μετά την, θέση, μετά την υλοποίηση της συνθήκης της ε, ε, Λισαβόνας σε ε, παιδεία όπως η ε, δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν και τη δική σας επιτροπή. Τον Μάρτιο του 2014 οργανώσαμε μία κρόαση και ο Ζων Κλώτ Τρισέ, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο κύριος ε, Μάρτιν Κέρε από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετέσχουν και μετά από τις, από εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ταξιδέψαμε στις Βρυξέλλες και συζητήσαμε με βασικούς φορεί από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Απασχόλησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με εκπροσώπους του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η έκθεσή μου βασίζεται στις βασικές αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε ορισμένου τομεί προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε και υψηλότερη προστασία ε, σε σχέση με ε, τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια έχει και δικά της σημεία στα οποία εστιάζει. Το Μάρτιο του 2014 η έκθεση για την ενίσχυση του κράτους δικαίου είναι ένα παράδειγμα ενός μηχανισμού για την αντίδραση σε απειλές ε, στο κράτος δικαίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έπρεπε να υπάρχει συντονισμός με το κεκτημένο του Συμβουλίου της Ευρώπης και όχι μόνο αυτά τα οποία, και να μην γίνονται μόνο αυτά τα οποία προτείνονται από την Επιτροπή στο προήμιο. Θα πρέπει νομίζω όλα τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, να λαμβάνονται υπόψη σε τέτοιου είδους μηχανισμούς ε, και ε, δηλαδή δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκθέσει τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκθέσει τη επιτροπή παρακολούθηση των Εργασιών τη κοινοβουλευτική συνέλευση. αρκετές φορές ε, η Κοινοβουλευτική ε, Συνέλευση έχει εκφράσει τις ανησυχίες της για την επικάλυψη εργασιών. Το 2010 είχε τεθεί ένα θέμα τελευταία φορά όταν ο κύριος Σασίλοβιτς από την Λετωνία είχε κάνει μια έκθεση ε, και ένα ψήφισμα ανέφερε ακριβώς αυτό ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η επικάλυψη των εργασιών και από τον Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Επίσης, όταν ε, σκεφτούμε την κατανομή κονδυλίων σε διάφορους οργανισμούς ε, και για την ε, έρευνα και ανταλλαγή απόψεων, θα πρέπει να αποφεύγουμε την επικάλυψη. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να έχουν ένα διαρθρωμένο διάλογο και να μην υπάρχει επικάλυψη γνωρίζοντας ότι η χρηματοδότηση ούτως ή άλλως είναι ε, μικρή. Θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνουμε τα μέτρα μας ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη. Ε, αναφέρομαι στην έκθεσή μου και για την ε, προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην απόφαση του Δεκεμβρίου του 2014 Το ύφος ε, της γνωμοδότησης ήδη έχει συζητηθεί και έχει σχολιαστεί ε, και πολλοί έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους. Φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια στην ε, οριστικοποίηση των ε, συζητήσεων και φαίνεται ότι η τελική συμφωνία θα είναι ε, μακροχρόνια αν όχι αδύνατη. Ελπίζω ότι οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρουν έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τίθενται οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας επίσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ε, τις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αποφάσεις αυτών των οργάνων επιβάλλουν μέτρα λιτότητα σε κάποια μέλη της Ευρωζώνης καθοδηγούμενα ε, από, το ότι, ε, από θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων το, το συμπέρασμά μου λέει ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και έλλειψη δημοκρατικής διαδικασίας για ορισμένες τέτοιες αποφάσεις. Έχει ε, εξεταστεί το θέμα αυτό και από άλλους φορείς της ε, κοινοβουλευτικής διάσκεψης και δεν ήθελα ε, να επαναλάβω αυτά τα οποία ήδη έχουν υποθεί αλλού. Εγκρίθηκε τέλος μετά την έκθεσή μου το ψήφισμα 2041 που ζητά από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να δώσουν άμεση προτεραιότητα σε αυτό το θέμα. Επίσης, καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει με διαρθρωμένο τρόπο τη συνεργασία της με το Συμβούλιο της Ευρώπης και να χρησιμοποιήσει την εμπειρία που έχει το Συμβούλιο της Ευρώπης και την ε, εμπειρογνωμοσύνη του. Όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το Μηχανισμό και το Κράτος Δικαίου, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ήταν τη γνώμη ότι θα πρέπει να ενημερώνονται για όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία που έχει αναπτύξει το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Τέλο, η άποψη τη Κοινοβουλευτική Διάσκεψη είναι ότι θα πρέπει να εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα σχέδια νόμων της, ε, ούτως ώστε να είναι συμβατά με το χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό πιστεύω ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εσάς που είστε εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως επίσης και το προσωπικό του Κοινοβουλίου και την νομική υπηρεσία. οι επιπτώσεις των σχεδίων νομοθετικών κειμένων στα θεμελιώδη δικαιώματα εξετάζονται όπως επίσης εξετάζονται και τα θέματα των τροπολογιών που είναι σημαντικό τμήμα της ε, νομοθετικής διαδικασίας. Θα ήθελα λοιπόν και τη δική σας ε, άποψη όσον αφορά και τις τροπολογίες ε, στις Βρυξέλλες είχα συναντήσει κάποιους συνομιλητές μου είχαν πει ότι δεν έχουν επαρκείς πόρους οι νομικές υπηρεσίες για να μπορούν να εξετάζουν όλες τις προτινόμενες τροπολογίες δεν έχουν τους πόρους για να εξετάσουν τις επιπτώσεις που θα είχε κάτι τέτοιο επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων Τέλος, η συνέλευση επανέλαβε την έκκλησή της προς τα κράτη-μέλη να ε, εξετάσουν ε, την ε, προσχώρηση στη Σύμβαση Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θα πρέπει οι σχετικές συζητήσεις να αρχίσουν εκ νέου το συντομότερο δυνατόν και προτείνεται να γίνει και μία μελέτη ε, για να διατυπωθεί ένας κατάλογος κριτηρίων, ούτω ώστε μέτρα λιτότητας που τυχόν προτείνονται να μην έχουν επίπτωση στα κοινωνικο-οικονομικά δικαιώματα. Και η Επιτροπή Υπουργών ε, θα υποβάλει τις απόψεις της στην ε, κοινοβουλευτική διάσκεψη. Κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι η συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Συμβουλίου τη Ευρώπη που βασίζεται σε ε, μια συμφωνία του 2007 παραμένει σε ισχύ και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να αποφεύγουμε την επικάλυψη των εργασιών μας. Επίσης, ε, ελπίζω ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. και οι νομοθέτες θα πρέπει να φροντίζουν η προτινόμενη νομοθεσία να μην έχει επιπτώσεις, ε, αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, σας ζητώ να εξετάσετε τις συστάσεις ε, που υπάρχουν στο ψήφισμα 2041 και να τα λάβετε υπόψη σας στο έργο της Επιτροπής σας. Καθώς και στην εκπόνηση νομοθετικού έργου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να διατηρήσουμε υψηλά ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κοινό μας ευρωπαϊκό χώρο. Ιδίω η ιδέα της ενίσχυσης, της παρακολούθησης, της στήριξης των κριτηρίων της Κοπενχάγης από τα κράτη-μέλη είναι μια ιδέα που καταρχήν χαιρετίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και οποιαδήποτε πρωτοβουλία σε αυτό τον τομέα θα πρέπει να είναι αντικείμενο συντονισμού με το Συμβούλιο της Ευρώπης για να αποφεύγουμε περιττή επικάλυψη. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη εκτίμησή μου για τη γραμματεία σας που συνάντησα κατά την επίσκεψή μου τον Ιούνιο, γιατί τότε δεν είχα συναντήσει βουλευτές καθώς δεν υπήρχαν ε, συνεδριάσεις μετά τις εκλογές και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία σας, ε, για, τις σα, για τη βοήθεια κατά την, που μου έδωσαν κατά την σύνταξη τη εκθεσή μου. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και περιμένω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μακναμάρα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Ένα συνάδελφος επιθυμεί να πάρει το λόγο. Η κυρία Σίπελα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Μακναμάρα Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας, που νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι και αυτή η έκθεση και άλλες εκθέσεις τις οποίες λαμβάνουμε μας τρομάζουν, γιατί νομίζουμε ότι είναι όλα εντάξει στην Ευρώπη και Συνήθως ασκούμε κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε άλλες ε, περιοχές και ξεχνάμε ότι και σε εμά ε, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα. Είναι λοιπόν πολύ χρήσιμο το να κρατάμε ένα καθρέφτη μπροστά μας, να μπορούμε να βλέπουμε και το τι συμβαίνει στη δική μας την αυλή. Και ε, αναφέρονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένα κράτη-μέλη και για προβλήματα συντονισμού και εποπτείας ε, σχετικά με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές έχει ζητήσει να γίνεται μια τέτοια παρακολούθηση των κριτηρίων της Κοπενχάγης. Ε, ε, ξέρω ότι από την πλευρά της Επιτροπής ε, αλλά και από άλλους ε, τίθεται το ερώτημα του ποια είναι τα κριτήρια τα οποία θα θέσουμε ε, σε αυτήν την παρακολούθηση. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι τα κριτήρια και να καταλήξουμε σε κάποια έκθεση για όλα τα κράτη-μέλη. Φοβούμαι ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμη. Θυμάμαι από την περασμένη θητεία είχαμε ζητήσει από την Επιτροπή τότε να γίνει μια παρακολούθηση των επιπτώσεων που δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι, τότε, μέχρι τώρα. Φοβάμαι ότι αυτό δεν είναι απλώς θέμα έλλειψης προσωπικού, αλλά ίσως υπάρχει και έλλειψη πολιτικής βούλησης σε ορισμένα σημεία. σε άλλες περιπτώσεις ε, άλλα θέματα διεκπεραιώνονται πάρα πολύ γρήγορα. Ίσως λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο εμποδίζει τα συγκεκριμένα θέματα. Έκανα αυτές τις εισαγωγικές ε, παρατηρήσεις, αλλά έχω και κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Η πρώτη μου ερώτηση είναι αν υπάρχουν ήδη επαφές ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναφέρατε τον οργανισμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά έχετε επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς διαφρώνεται η συνεργασία με το Συμβουλίο της Ευρώπης. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα δικά σας κριτήρια όταν εξετάζετε την τήρηση των θεμελιωδών αξιών. Και όσον αφορά τη συστηματική παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα με ενδιέφερε αν θα μπορούσατε να μας πείτε εσείς αν, έχει αυξηθ, αν έχουν αυξηθεί αυτές οι παραβιάσεις τα τελευταία χρόνια και αν από τη δική σας εμπειρία παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, γίνονται σε πολλά κράτη-μέλη και αν έχουν προκύψει και κάποιοι τομείς τα τελευταία χρόνια όπου έχετε δει ότι ε, παρατηρούνται ιδιαίτερως ε, παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή αν υπάρχουν άλλοι τομείς στους οποίους δεν υπάρχουν παραβιάσεις. Ευχαριστούμε κυρία Τζίπερ. και κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Υποστηρίζω αυτά που μας είπε μόλις τώρα η κυρία Σίπελτ. Και εγώ ενδιαφέρομαι για το θέμα. Το πώς η λιτότητα επηρεάζει την κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είμαι μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης του Ευρωκοινοβουλίου και είναι κάτι που μας απασχολεί. Και σε εκθέσεις του προηγουμένου Κοινοβουλίου αναφέρεται το θέμα όπως αντίκτυπος των αποφάσεων της Τρόικα. Βλέπουμε ποια είναι η σχέση μεταξύ των αποφάσεων που λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι χρηματοσωτικής φύσεως, και τι αντίκτυπο έχουν από την άλλη πλευρά σε εθνικό επίπεδο. Είναι τομεί πολύ συχνά εθνική αρμοδιότητα, όπω πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κλπ. κλπ. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε κατά πόσο υπάρχουν κάποιες ιδέες σχετικά με το πώς μπορούμε να πετύχουμε καλύτερο συντονισμό. Συντονισμό με το Συμβούλιο της Ευρώπης που εκεί αντιπροσωπεύονται πολύ περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια και σχετική τους διάσταση. Υπάρχουν ιδέες που θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στη δική μας αξιολόγηση των προγραμμάτων μας των εξαμήνων όταν εξετάζουμε τις αιτήσιες συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Εθνικές Πολιτικές όπου υπογραμμίζονται και αναφύονται τέτοια θέματα. Μήπως μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα. Αναφερθήκατε και στα κριτήρια της Κοπενχάγης και πώς εφαρμόζονται. Είναι κάτι που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Το βασικό στοιχείο επιρροής είναι πριν την προσχώρηση μιας χώρας. Και μετά θεωρείται σαν δεδομένο ότι η χώρα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά έχουμε πλήρη επίγνωση το ότι υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, πώς μπορούμε το όλο θέμα να το προσεγγίσουμε και να το παρακολουθήσουμε. Σε ενδιαφέρει πολύ. Να μην λέμε στον υπόλοιπο κόσμο τι πρέπει να κάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά να ασκούμε και αυτοκριτική σχετικά με το τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Ευχαριστώ, Τζέιν Λάμπερτ. Ο κ. Χρυσόγονος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά την ανταπόκριση, πώς θα ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οικονομική κρίση. Η έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης σωστά υπογραμμίζει ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται και τη σχετική διαδικασία. Και υπάρχει και έλλειψη ελέγχου εκείνων που παίρνουν τι αποφάσεις. Πρέπει να δούμε ότι δυόμιση και τρία χρόνια μετά την δημοσίευση σειράς αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κοινωνικά δικαιώματα που θεώρησε θεωρητικά την Ελλάδα και πρακτικά την ε, Τρόικα ότι παραβιάζουν αρκετές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Χάρτας λόγω υθετηθέτων μέτρων που υθετήθηκαν λόγω λιτότητας. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε τίποτα για να σταματήσει το πρόβλημα και οι παραβιάσεις Απολύτως τίποτα δεν έγινε. Αντίθετα μάλιστα. Είναι εξωφρενικό και εξοργιστικό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαιτούν τώρα η νέα ελληνική κυβέρνηση που έχει λαϊκή εντολή για να θέσει τέρμα στην λιτότητα να λησμονήσει η κυβέρνηση την εντολή και να προχωρήσει περαιτέρω παραβιάζοντα την Ευρωπαϊκή Χάρτα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Παραδείγματο χάρη νομιμοποιώντα τι μαζικέ απολύσει εργαζομένων από του εργοδότε παρά το άρθρο 4 τη Χάρτα. Ακόμα πιο εξωφρενικό και εξοργιστικό είναι ότι πολλά από αυτά τα αιτήματα δεν έχουν καμία σχέση με την οικονομική σταθερότητα ή οδήποτε οικονομικό κέρδος και εξυπηρετούν απλώς την αύξηση των κερδών των ε, κεφαλαίων, του μεγάλου κεφαλαίου. Άρα κάποιος πρέπει να διερωτηθεί. Η λιτότητα είναι ένα μέσο καταπολεμήσεως της χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή όπως αλλιώς αποκληθεί ή η υπερχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι ένα μέσο προς τον σκοπό που είναι αυτή καθεαυτή η λιτότητα. Διότι η λιτότητα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το μερίδιο του κεφαλαίου στον αφορά το εθνικό εισόδημα μιας χώρας αυξάνεται εις βάρος των εργαζομένων. Και ίσως η ελίτ, η ευρωπαϊκή, αυτό έχει σαν στόχο τελικά. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ερώτησή μου προς τον κύριο Μακναμάρα συμπληρώνει εκείνη του συναδέλφου του κυρίου Χρυσογόνου. Αυτό που ήθελα να είναι ακριβώς τι, τι σημαίνει να υπάρχει, ένα, να υπάρχει ευρωπαϊκό δικαίωμα όταν βλέπουμε από την άποψη του Συμβουλίου ε, της Ευρώπης και από την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σας ρωτώ αυτό διότι το Συμβούλιο της Ευρώπης σε δύο συνελεύσεις το 2012 και το 2014 σαφώς κατήγγειλε την παραβίαση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων λόγω των πολιτικών λιτότητας σε δύο ψηφίσματα τα οποία επενθυμίστηκαν σωστά από το συνάδελφό μου τον κύριο Χρυσόγονο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αυτή την τοποθέτηση από την έποψη του δικαίου αυτού καθεαυτού. Δηλαδή η απάντηση που δόθηκε σε μια ερώτηση όσον αφορά τις συνέπειες των πολιτικών λιτότητας επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η απάντηση που δόθηκε από τον Επίτροπο Κατάινεν εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Σώματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν η εξή. Ότι κατά κάποια έννοια ο Ευρωπαϊκός νόμος, το κράτος δικαίου, το rule of law που εδράζεται επί της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων αναστέλλεται στην περίπτωση της Ελλάδας διότι η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα κρατικού χρέους που θα πρέπει να επιληθεί με τους ίδιους τους πιστωτές της. Αυτό που σας ρωτώ λοιπόν είναι, εσείς καταγγέλλετε τις συνέπειες επί των δικαιωμάτων από πλευράς πολιτικής λιτότητας που δεν βασίζονται οι πολιτικές λιτότητες σε, κανένα δικαίωμα, σε κανένα ιδέα δικαίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει άλλη αντίληψη. Είναι αυτό ένα από τα προβλήματα λόγω των οποίων δεν καταφέρνουμε δεν μπορεί να προσχωρήσει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο της ε, Ευρώπης. Ευχαριστώ κυρία Σπινέλη. Τώρα θα δώσω το λόγο στον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Μακναμάρα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να διατρέξω όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Σίπελ και για τον τρόπο με τον οποίο με στηρίξατε, συμφωνήσατε με αυτά που είπα, σε αυτά που είπα. Ρωτάτε, ποια είναι η βάση όπου εδράζονται κάποια δικαιώματα ε, και πώς αξιολογούμε τα δικαιώματα αυτά. Καταρχά είναι τα δικαιώματα τα οποία βασίζονται στη Χάρτα Θεμελιών Δικαιωμάτων, στην Συνθήκη τη Λισαβόνα, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που έχει την ίδια εντομική ισχύ με τι Ευρωπαϊκέ Συνθήκε και τη Συνθήκη τη Λισαβόνα. Και υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα που παίζει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη των δικαιωμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο. Μιλήσατε για τις απειλέ στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη. Υπάρχουν διάφορες απειλές και υπάρχουν και διάφορες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κάθε κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε απλώς τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να δείτε ότι έχω δίκιο. Για τις συστημικές απειλές. Το θέμα των εθνικών μειονοτήτων στις βαλτικές χώρες. οι Βαλτικέ χώρε είπαν ότι δεν θα αντιμετωπίσουν τι μειονότητες, αλλά τα προβλήματα των παραβιάσεων των, ε, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων μετά την ε, προσχώρησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δέκα χρόνια μετά την προσχώρησή του, τα προβλήματα σεβασμού των ε, εθνοτικών αυτομειονοτήτων και τη προσχώρησή του, τη απόκτηση κάποια ηθαγένεια, δεν έχουν λυθεί. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετωπίζουν προβλήματα σεβασμού των δικαιωμάτων των ετών των άσυλων και την αποσύνδεση. Κοιτάξτε, όταν γίνεται λόγος ε, για αυτά τα θέματα, εγώ ξέρω ότι ανακύπτουν πάρα πολλές φορές τα προβλήματα των ετούντων άσυλο. Ε, σας μιλάω και ως Ιρλανδός ε, ε, βουλευτής. Ε, μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και για άσυλο τα, και τα συζητάμε χωριστά τα αποσυνδέουμε. Λες και δεν συγκλίνουν, λες και δεν συνδέονται. Επίσης υπάρχει απειλή, μια άλλη συστημική απειλή, ε, απειλή στο κράτος δικαίου. Και ο διαχωρισμός εξουσιών α, στα κράτη-μέλη. Παραδείγματος χάρη ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Το δικαστικό σώμα ε, δέχεται πάρα πολλές απειλές. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός να αντιδράσουμε σε αυτές τις ε, αλλεπάλληλες συστημικές απειλές. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μηχανισμό που θα αντιμετωπίσει κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευτυχώς έχουμε δικαστήρια γι' αυτό. Και έχουν γίνει πάρα πολλά για να μεταρρυθμιστούν τα δικαστήρια, ο τρόπος που λειτουργούν, ε, να σταματήσει η συσσόρευση υποθέσεων, η καθυστέρηση της διεκπαιρέως των υποθέσεων κτλ. Ε, και αυτή είναι η αντίδραση των πολιτικών στις ε, συστημικές απειλές. Τώρα, το κατά πόσο τις αγνοούν, ακριβώς αυτό αντιμετωπίζει η έκθεση. Η κυρία Λάμπερτς τώρα. Η ερώτησή σας αφορούσε το αν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχει μία. Ο κύριος ε, Jean-Claude ε, Trichet παρέστησε μια συνάντηση της Επιτροπής και εξέφρασε την απόψή του για τις δράσεις που αναλαμβάνονται και συνέκρινε είπε μάλιστα ότι η θέση του είναι σαν να είναι μέσα στο πιλωτήριο ενός αεροπλάνου το οποίο ταξιδεύει προς ένα άγνωθο προορισμό ε, όταν, ε, μετά την περίοδο που κατέρευσαν οι τράπεζες. Κατά την άποψή του, τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι ανεξάρτητα από την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ ε, θεσπίζει την νομισματική πολιτική ανεξάρτητα, έτσι, χωρίς πιέσεις. Γιατί αυτό το προβλέπει η συνθήκη, οι συνθήκες. Και τώρα ε, επιπλέον πρέπει να πούμε ότι τα περισσοτερα κατημέλη έχουν ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες. Η ΕΚΤ θέτει τα επιτόκια λαμβάνοντας υπόψη μόνο τον πληθωρισμό και όχι να λάβει υπόψη τη τα θέματα απασχόλησης όπως το κάνει η ΦΕΔ στην Αμερική. Όλα τα θεσμικά όργανα ε, δεσμεύονται από τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τα μέτρα που έχει. Και η Χάρτα μιλάει για το δικαίωμα στην εργασία. Πάει πολύ πιο πέρα από άλλα έγγραφα. Κοίταξα την ε, γαλλική και αγγλική εκδοχή της χάρτας και λέει κατηγορηματικά στο άρθρο 15 ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν. Κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την ελευθερία να αναζητήσει εργασία για να εργαστεί. Έχει την ελευθερία να αναζητήσει εργασία ή την ελευθερία να εργαστεί. Επίτηδες τα μπλέξανε λίγο αυτά τα θέματα ε, στη χάρτα όταν την συντάξανε. Θα ήταν πάντως περίεργο η ΕΚΤ να αγνοήσει εντελώς ε, τις επιπτώσεις των μέτρων της στο δικαίωμα εξέβρασης εργασίας στην Ευρώπη. Ίσως θα πρέπει και η ΕΚΤ να, προσκαλ... να καλείται να συνεργάζεται πιο στενά όταν ε, αναπτύσσει τις πολιτικές της, ούτως ώστε να βλέπουμε και τις επιπτώσεις των πολιτικών της στα κοινωνικο-οικονομικά δικαιώματα. Έχουμε αυτή την ε, πολιτική ορθοδοξία στην ε, Ευρώπη. Ότι έχουμε από τη μία τα οικονομικά θέματα και από την άλλη τα κοινωνικά δικαιώματα. Και αυτό συνεισφέρει στην έλλειψη σεβασμού για την επίπτωση των ε, μέτρων για την επίπτωση των μέτρων λιτότητας στις, σε κοινωνικά και οικονομικά θέματα. Κύριε Χρυσόγονε, παρακολούθησα με ενδιαφέρον όλα όσα συμβαίνουν στην ε, Ελλάδα. Και ως Ιρλανδός βουλευτής ε, μίλησα για τα θέματα της διάσωσης και έχω τεράστια συμπόνια και κατανόηση για τη θέση των ε, Ελλήνων ερετών αρχόντων. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ της Ιρλανδίας και αυτών που προτείνονται για την Ελλάδα. Ως μέλος του Εργατικού Κόμματος, που ανήκει στους, στην ομάδα των σοσιαλιστών, υποστήριξα μέτρα που δεν φανταζόμουν ποτέ παλιά ότι θα μπορούσα να υποστηρίξω. Η Ιρλανδία όμως σε μεγαλύτερο βαθμό από την Ελλάδα μπόρεσε να επιλέξει τα μέτρα που εφάρμοσε Νομίζω, ότι δεν είμαι εμπειρογνώμων για τα θέματα της Ελλάδας, ότι η Ελλάδα δεν έχει αυτή την επιλογή καθόλου. Πολλά μέτρα επιβλήθηκαν στην Ελλάδα. Αλλά έγιναν και πολύ δύσκολες επιλογές, πρέπει να το πω αυτό, στην Ιρλανδία. Δύσκολες αποφάσεις που ελήφθησαν. Σε καμία περίπτωση δεν εννοώ ότι όταν ε, μια χώρα αντιμετωπίζει κρίση δημοσίου χρέους δεν θα υπάρξουν δυσκολίες. Ο Τρισέ είπε ότι έχουμε δύο εναλλακτικέ. Είτε ε, ευθυγραμμίζουμε τις δαπάνες με τα εισοδήματα ή θα μειώσουμε πάρα πολύ τις ε, δαπάνες. Το κάναμε αυτό στην Ιρλανδία. Αλλά αυτό δεν επηρέασε τα κοινωνικο-οικονομικά δικαιώματα, όπως παραδείγματος χάρη το δικαίωμα στις ε, συλλογικές συμβάσεις που αναφέρατε. Ε, και δεν είχαμε παραβιάσεις αυτού του δικαιώματος, ενώ στην Ελλάδα είχαμε. Η κυρία Σπινέλη, από την Ισπανία, λέει από την Ιταλία. Συγγνώμη. Λέμε για την έννοια που έχει ο καθένα για το δίκαιο, για το πώ αντιλαμβάνεται κανένα το δίκαιο. Υπάρχει μια κάποια ορθοδοξία στην Ευρώπη που διαφοροποιεί τα κοινωνικο-οικονομικά δικαιώματα και τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και θεωρείται ότι τα κοινωνικο-οικονομικά είναι λιγότερο σημαντικά. Η προσωπική μου άποψη ποια είναι. Ότι πρέπει να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. και οι υπερεθνικές οντότητες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ε, όταν δεν είχε την δημοκρατική νομιμότητα που έχει τώρα, από πού αποκτούσε την ε, νομιμότητά της, από την ικανότητά της που είχε να διεκδικεί αυτά τα δικαιώματα. Όταν τα υποσκάπτει, όταν δεν τα ε, προστατεύει τα δικαιώματα χάνει αυτή την νομιμότητα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μακναμάρα, ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας για τις ενδιαφέρουσες σκέψεις σας και για τις δοθείς σας πληροφορίες. Είναι ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας που θα πρέπει να συνεχιστεί. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Και σας εύχομαι καλή συνέχεια στη δουλειά σας θα πρέπει να διακόψουμε τη συνεδρίασή μας για ένα τέταρτο διότι η κυρία Βίξτρομ η είναι εδώ αλλά υποθέτω ότι δεν έχουμε τους άλλους προσκεκλημένους μας που ίσως ζητήσουν να παρέμβουν στην συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να περιμένουμε μέχρι... Είναι εδώ? Αν δεν είναι εδώ πρέπει να περιμένουμε. Αν είναι εδώ μπορεί να συνεχίσουμε. Δέκα λεπτά διάλειμμα. Yeah, ja,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

So, colleagues, uh, we, we could continue with our... Ας συνεχίσουμε με τη συνεδρίασή μας, την απογευματινή. Ask everybody to... Λοιπόν, παρακαλώ, καθίστε. Let us continue the meeting. Ας συνεχίσουμε. θα έχουμε αρκετούς ενδιαφερόμενους απόψε. Θα περιμένω μέχρι ότου καταφτάσει η Σεσίλια και καθίσει. Στο σημείο 6 λοιπόν της ημερήσιας διάταξής μας έχουμε το θέμα της, του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο να εξετάσει ε, το, ε, την αίτηση για διεθνή προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ζητώ την κυρία Βίξτρομ που είχε ασχοληθεί με τον κανονισμό του Δουβλίνου επί Μακρόν να κάνει μια εισαγωγή. Μετά από αυτό έχουμε καλέσει κάποιους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους να προβούν σε σύντομη ε, δήλωση όσον αφορά τα απορίσματά τους αν θεωρούν ότι θα πρέπει να συντάξουμε κάποιο έγγραφο τοποθέτηση στον αφορά το νομοθέτημα ή αν αφορά μόνο ένα άρθρο, το άρθρο 8 του κανονισμού και μια παράγραφο αυτής. Πρώτα να σας δώσω το λόγο κυρία Βίκστρομ και μετά θα ακούσουμε τους προσκεκλημένους μας και τους σκιώδεις εισηγητές. Η κυρία Βίκστρομ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Διατρέχω τον κίνδυνο από ό,τι καταλαβαίνω να επαναλάβω αυτά που έχω πει, αλλά εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συνοψίσουμε το ιστορικό της εκθέσεως. Ξεκίνησε στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου, ήμουν εισηγήτρια για την ανδιατύπωση του κανονισμού του Δουβλίνου που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2013. Όμως υπήρχε μία παράγραφος ενός άρθρου που δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε, το άρθρο 8, παράγραφος 4, που αποφάσισε ποιο κράτος μέλος έχει την ευθύνη για αίτηση ασύλου όσον αφορά ασυνόδευτους ανήλικους. Ο παλαιός κανονισμός του Δουβλίνου δεν ήταν καθόλου σαφής από αυτού. Δεν διευκρίνεζε αν είναι το, η πρώτη ή πλέον πρόσφατη αίτηση εκείνη στην οποία εφαρμόζεται ο Γενικός Κανόνας. Όταν ο προηγούμενο κανονισμό του Δουβλίνου ήταν αυτό που ίσχυε, ερμηνευόταν από τα περισσότερα κράτη-μέλη ω εξή. Ότι και ασυνόδευτοι ανήλικοι θα μπορούσαν να ε, επιστρέψουν στο κράτο μέλο από το οποίο, ε, στο οποίο κατέφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχήν ο ασυνόδευτος ανήλικος. Στην αδιατύπωση του κανονισμού του Δουβλίνου όλα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν σε διασαφήνιση του όρου, αλλά, και αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε στο πώς θα πετύχουμε αυτό το στόχο και πώς θα ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ήθελαν να διευκρινιστεί ότι το κράτος εκείνο το οποίο ο ανήλικος είχε υποβάλει την πλέον πρόσφατη αίτηση που έχει την ευθύνη. Το Συμβούλιο όμως επέμενε ότι πρέπει να είναι η χώρα εκείνη της υποβολής της πρώτης αιτήσεως και δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε. Την εποχή των διαπραγματεύσεων εκρεμούσε υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πάνω στο ίδιο θέμα. Και εφόσον δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε, αποφασίσουμε να αφήσουμε το κείμενο είχε στον παλιό κανονισμό, αλλά προσθέσαμε υπό την προϋπόθεση ότι είναι προς το καλύτερο συμφέρον του ανηλίκου. Και κάναμε κάτι άκρος ασύνηθες, καταφέραμε να προβούμε σε κοινή δήλωση που υποστήριξαν και τα τρία θεσμικά όργανα και δηλώναμε ότι από τη στιγμή που θα υπήρχε απόφαση του δικαστηρίου επ' αυτού, η Ευρωπαϊκή Επίτροπη θα έπρεπε να ξανανοίξει τη συγκεκριμένη παράγραφο του κανονισμού του Δουβλίνου και να επιστρέψει με πρόταση η οποία θα αντικατόπτριζε απολύτως την απόφαση του δικαστηρίου. Και τέλος η απόφαση ελήφθη τον Ιούνιο του 2013 πριν την έγκριση του κανονισμού του Δουβλίνου. Η απόφαση ευθυγραμμιζόταν ε, με την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, δηλαδή ότι πάντα θα πρέπει να αποφευχθούν ε, α, μη απαραίτητε μεταφορές των ανηλίκων και το κράτος υπεύθυνο για το συνόδευτο ανήλικο θα πρέπει να είναι το κράτος εκείνο το οποίο είναι παρόν το ανήλικο άτομο. Πρώτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει το κείμενο, δεόντως και τον Ιούνιο του 2014, ένα χρόνο μετά, έκανε την πρότασή της και οι συνομοθέτες θα πρέπει να ενστερνιστούν αυτή την αλλαγή. Είναι αναμφισβήτητο ότι θα πρέπει πάντα να δρούμε προς το βέλτιστο όφελος του παιδιού που είναι κάτι που αναφέρεται και στο άρθρο 24 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η απόφαση του δικαστηρίου επίσης αναφέρει ότι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα και συνεπώς θα πρέπει κατά κανόνα να μην μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος. Εγώ, όπως και συνάδελφοι, καλωσορίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιστεύω ότι εγκατοπτρίζει άριστα την απόφαση του δικαστηρίου, όπως συμφωνήσαμε και στην διακήρυξη, στη δήλωση και αντικατοπτρίζει και την Αθνική Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αδιατύπωση του κανονισμού του Δουβλίνου. Εν γέννη λοιπόν, απλό είναι το καθήκον και ο στόχο μα και παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι δύσκολο ο στόχο. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε αυτό το άθρο με την απόφαση του δικαστηρίου διότι συμφώνησα να το κάνω αυτό και τα τι θεσμικά όργανα στην κοινή αυτή δήλωση. Εγώ παρουσίασα το σχέδιο εκθέσεώς μου τον Ιανουάριο και εκεί ε, υποστήριξα πλήρως την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εφόσον αφορά μόνο μία μικρή παράγραφο ενός άρθρου ε, δεν είδα να υπάρχει ανάγκη να επιφέρουμε κάποιες αλλαγές. Και δεν έχω εισαγάγει καμία αλλαγή, απολύτως καμία αλλαγή στο διατακτικό του κειμένου, απλώς προβαίνω σε κάποιες ε, διασαφηνίσεις στα αιτιολογικά, στην αιτιολογική έκθεση. Και οι λέξεις που χρησιμοποιώ αντεγράφησαν από την απόσταση του δικαστηρίου και τη γνωμοδότηση του Γενικού ε, η εισαγγελέα και αυτά σύμφωνα με αυτά που είπαμε. Και ο βασικός κανόνας ποιος είναι, ότι το κράτος μέλος όπου είναι παρόν το ανήλικο άτομο θα πρέπει να μεριμνήσει για την αίτηση ασύλου του ανηλίκου. Όμως, η βασική επικρατούσα αρχή ποια είναι, το καλύτερο συμφέρον του ανηλίκου. Και δεν αποκλείεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ενδεχομένως, θα μπορούσε να είναι προς το καλύτερο όφελος του ανηλίκου να μεταφερθεί. Αλλά αυτό θα πρέπει να εδράζεται επί ατομικής αξιολογήσεως του καλύτερου συμφέροντος του ανηλίκου και αυτό θα πρέπει να γίνει πριν ληφθεί η αδίποτε απόφαση περί μεταφοράς αυτού. Το δικαστήριο λοιπόν αναφέρει τρεις αρχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη και με την εξή σειρά. Πρώτα απ' όλα, το καλύτερο συμφέρον του ανηλίκου. Δεύτερον, να μην υπάρχει ε, περιττή μεταφορά και τρίτον, ταχεία πρόσβαση στη διαδικασία χορηγήσεως ασύλου. Ε, ανησυχώ πάρα πολύ ε, για την θέση του Συμβουλίου, διότι ανοίγεται για μεταφορά ανηλίκων αν η διαδικασία ήδη έχει ξεκινήσει σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, διότι υπολείπεται κατά πολύ τη αποφάση του δικαστηρίου που αναφέρεται στην αρχή σύμφωνα με την οποία ε, το κάτω μέλος στο οποίο είναι παρόν το ανήλικο άτομο είναι υπεύθυνο για την αίτηση ασύλου και αναμφισβήτητα ανοίγει ε, το δρόμο για περιτές μεταφορές και συνεπώς παρατείνει την όλη διαδικασία. Ξέρουμε ότι οι μεταφορές είναι χρονοβόρες, είναι πιο χρονοβόρες ε, από το να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία ασύλου. Άρα είναι βασικό, σημαντικό και πάντα ήταν έτσι σε όλη τη διαδικασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σεβαστούμε την ε, δήλωση που ε, υπέγραψαν και τα τρία θεσμικά όργανα άρα πλήρως ευθυγραμμιζόμεθα με την απόφαση του ε, δικαστηρίου. Επουδενή σε καμία περίσταση δεν θα έπρεπε να αποδεχτούμε οδήποτε κείμενο το οποίο θα υπολείπεται της αποφάσεως και σας παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι αναφερόμαστε σε ευάλωτα παιδιά και νομίζω ότι όλοι κατανοούμε και βλέπουμε γιατί χρειάζεται αυτό να λάβουμε κάθε προφύλαξη για να τα προστατεύσουμε τα παιδιά. Καλωσορίζω λοιπόν τις τροπολογίες που υπευλήθησαν από συναδέλφους διότι όλες οι τροπολογίες ακολουθούν αυτή την γραμμή και σέβονται αυτό το πνεύμα. Θα πρέπει να κρατήσουμε το κείμενο πολύ ξεκάθαρο, όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται, αλλά όσον αφορά το περιεχόμενο, όλοι είμαστε συντονισμένοι και προσβλέπω σε λεπτομερέστερες συζητήσεις επί της οδηγίας με όλους τους σκιώδεις ηγητές σε επικείμενη συνεδρίαση των σκιωδών. Και χαίρομαι όλους ιδιαίτερο σήμερα διότι η Επιτροπή μας ε, δίνει τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους φορείς, ενδιαφερόμενους που κατάφεραν να βγουν από τα σανσέρ στο οποίο είχαν κολλήσει για κάποια λεπτά, να είναι εδώ διότι ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι με τα θέματα των ασυνόδευτων ανηλίκων και νομίζω ότι είναι σημαντικότατο για όλους μας έτσι να τους ακούσουμε για λίγο, να ακούσουμε τι έχουν να μοιραστούν μαζί μας όσον αφορά τα απορίσματά τους εκεί, στην πράξη, επιτόπου, στον πραγματικό κόσμο όταν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να αποτελέσει προστεθέμενη εξιά και για τις μελλοντικέ μας διαπραγματεύσεις να λάβουμε υπόψη αυτά που θα μας πούν και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του Συμβουλίου, όπως πάντα, και θέλω να ακούσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, Σεσίλια. Πριν δώσουμε το λόγο... Και πριν δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας, θα ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής να λάβει το λόγο. Uh- ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμφωνώ καταρχήν με την κυρία Βίξτρομ ότι αυτά τα οποία σας λέω τώρα εν μέρη τα έχουμε ξαναπεί για την τέταρτη συνάντηση για το θέμα αυτό νομίζω. Θα ήθελα όμως να τονίσω για άλλη μια φορά τον συγκεκριμένο κανόνα που έχει η Επιτροπή για το θέμα αυτό. Έχει λάβει εντολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και τα δύο θεσμικά όργανα μας ζήτησαν να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό Δουβλίνο 3 όπως είπε η κυρία Βίξτρομ για να αναθεωρηθεί το άρθρο 4 μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ε, ε, υπόθεση 1α. Θα ήθελα επίσης ε, ε, να πω ότι χαιρετίζουμε το σχέδιο έκθεση της κυρίας Βίξτρομ που φαίνεται ότι ε, υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχέδιο έκθεσης προτείνει την ε, τροποποίηση ενός, μιας αιτιολογικής σκέψης και την προσθήκη δύο νέων. Όπως ήδη είπα στην παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης, η Επιτροπή θα μπορούσε καταρχήν να υποστηρίξει τους στόχους, όμως ορισμένα θέματα απαιτούν συζητήσεις και διευκρινήσεις σε τεχνικό επίπεδο, ούτω ώστε να είναι σωστά από νομικής άποψης. Επίσης, θα ήθελα να πω, επειδή είχαμε την ευκαιρία να δούμε τις τροπολογίες, ότι το ίδιο μπορούμε να επαναλάβουμε και σχετικά με τις τροπολογίες στην έκθεση αυτή. Ορισμένε τροπολογίε φαίνεται ότι κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση. Παραδείγματο χάρη είναι τροπολογίε ε, που εισάγουν πιο σαφεί ε, διατάξει ε, για την προστασία του μείζωνο συμφέροντο του, του παιδιού. Αλλά όπω οι 18 και οι 19 μιλούν ε, για, τις, για τα αποτελεσματικά ε, ένδικα μέσα και κάποιες άλλες διαδικασίες ε, που έχουν σχέση με την οδηγία για την προστασία του ασύλου. Όλα αυτά όμως πρέπει να συζητηθούν και να αξιολογηθούν περαιτέρω όσον αφορά τις νομικές και τεχνικές πτυχές τους. Τρίτον τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτησε προσεκτικά όλες τις εκθέσεις των ενδιαφερομένων για το θέμα αυτό. Χαίρομαι που άκουσα ότι και οι ενδιαφερόμενοι υποστηρίζουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόσφατα κάναμε μια συνάντηση όπου το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Και θα ακούσω πολύ προσεκτικά τις δικές σας παρουσιάσεις σήμερα. Μήπως τυχόν υπάρχει κάτι νέο επιπλέον των συζητήσεων που ήδη έχουμε κάνει. Τέταρτο σημείο. Όπως και σε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις, θέλω να τονίσω κάτι που είναι τόσο σημαντικό που θέλω να το επαναλάβω η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδίω θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το μείζον συμφέρον του ανηλίκου είναι πάντοτε αυτό το οποίο την χάνει μεγαλύτερη ε, προσοχή σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην ε, υποθεση Μια 1α. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές νομικές απόψεις όσον αφορά την ερμηνεία. Τονίζουμε ότι είναι πολύ τεχνικό το θέμα και χρειάζονται συζητήσεις εμπειρογνωμόνων μεταξύ των νομοθετών και της Επιτροπής, αλλά θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση εδώ. Δηλαδή ότι ζητήθηκε από το δικαστήριο να ερμηνεύσει μια γενική διάταξη του κανονισμού Δουβλίνο 2 και επομένως δεν εξέτασε όλα τα πιθανά σενάρια τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν στην πράξη, στην πράξη για ε, ανηλίκους που υποβάλλουν αίτηση σε πολλά κράτη-μέλη. Και τονίζω ότι η ίδια η πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται σε κάποια σενάρια που δεν έχουν εξεταστεί άμεσα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πέμπτον, τονίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι μία ισορροπημένη συμβαστική λύση μεταξύ των νομοθετών και που αντικατοπτρίζει τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα τρία θεσμικά όργανα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το Δουβλίνο 3 είναι κάτι που θα μπορέσει σύντομα να εγκριθεί και ή δυνατόν πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι σημαντικό σημαντικό το να γίνει γρήγορα μια τέτοια ισορροπημένη συμφωνία, ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν υπόψη όσο δεν καλύτερα ε, τα συμφέροντα των ανηλίκων. Θα εξετάσει λοιπόν η Επιτροπή πολύ προσεκτικά τις θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τονίζω για άλλη μια φορά ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εμποδίσουμε ένα πολιτικό αδιέξοδο για το θέμα αυτό. Επί δύο χρόνια υπήρχε ένα πολιτικό αδιέξοδο και πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τα κενά και να μην εγκαταλείψουμε στην τύχη τους τους ασυνόδευτους ανηλίκους, αλλά να υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ευχαρίστως την χείρα βοηθείας και προς τα δύο θεσμικά όργανα στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και στρέφομαι στην ε, Προεδρία του Συμβουλίου. Θέλει να μας μιλήσει για τη γενική προσέγγιση που έχει ακολουθεί στο Συμβούλιο μέχρι τώρα. Ε, thank you, Madam. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Συμβούλιο έχει ε, επεξεργαστεί τις προτάσεις της Κομισιόν τις έχει εξετάσει και συμφωνεί με τα όσα είπε η μόνιμη Επιτροπή Εκπροσώπων της 5ης Φεβρουαρίου του 2015. Ακούσαμε αυτά που είπε η Κομισιόν, ότι θα πρέπει να ανοίξει ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο ώστε να υπάρξει συμφωνία επί της πρότασης, που είναι πολύ σημαντική. Το Συμβούλιο καθώς ε, ετοιμάζει τη θέση του για τον τριμερή διάλογο, πρέπει να πει ότι συμφωνεί πως το μείζον συμφέρον του παιδιού πρέπει να πριτανεύει σε όλες τις υποθέσεις. Αυτό είναι το σημείο αφετηρίας της πρότασης. Είναι σημαντικό, παράλληλα, να έχουμε σαφείς νομικούς κανόνες που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιθανά σενάρια. Όπως είπε και η Κομισιόν, οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν μπορούν να λάβουν υπόψη σε όλα τα πιθανά σενάρια. Το Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση της Κομισιόν και θεωρεί ότι οι ορισμένε προϋποθέσεις, οι μεταβιβάσεις αυτές μπορεί να είναι προς το συμφέρον των ασυνόδευτων ανηλίκων. Σε περίπτωση που οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πριν ε, υποβάλουν αίτηση για διεθνή προστασία που στα κράτη-μέλη που βρίσκονται παρόντα έχουν προηγουμένως υποβάλει άλλες αιτήσει σε άλλα κράτη-μέλη. Η μεταφορά μπορεί να είναι χρήσιμη σε αυτή την περίπτωση, η μεταβίβαση, γιατί ο ασυνόδευτος ανήλικος πρέπει να έχει ξεκάθαρη θέση για το δικαίωμά του για διεθνή προστασία. Όχι και όχι να περιμένει κατά πόσο θα ξεκινήσει η εξέταση της υπόθεσής του στο δεύτερο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται κιόλα. Το Συμβούλιο πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι προς το συμφέρον του παιδιού, προς το μείζον συμφέρον του παιδιού, να γίνει αυτή η μεταφορά. αλλά και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει μια ατομική εξέταση του μείζωνος συμφέροντος του συγκεκριμένου παιδιού. Όπως είπα και στην αρχή, ως Συμβούλιο περιμένουμε να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να έχουμε μια γρήγορη συμφωνία και γρήγορη οθέτηση της σημαντικής αυτής πρότασης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Έχουμε έξι ομιλητές. Σας καλώ όλους να περιοριστείτε σε τρία λεπτά. Δώσ' ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και συζήτηση. Θέλουμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της ε, ΥΠΑ της ε, Αρμοστίας, τον κύριο Φούνκεμαν. Την κυρία. την κυρία Φούνκεμαν. Ευχαριστώ την Επιτροπή Λίμπε για την ευκαιρία που μου δίνει να παρουσιάσω τις απόψεις ε, του, της αρμοστίας για το άρθρο 8.4. Το 6.1 του κανονισμού του Δουβλίνου θα πρέπει, λέει ότι θα πρέπει το συμφέρον του παιδιού να είναι το βασικό στοιχείο το οποίο ξεκινούν. Και μείζον συμφέρον αυτό σημαίνει το μισό συμφέρον. Δηλαδή, οποτεδήποτε λαμβάνουμε υπόψη την ε, μεταφορά, θα πρέπει να, να εξετάσουμε διάφορου παράγοντε, οι οποίοι περιγράφονται στο άρθρο 6.3 του κανονισμού ε, του Δουβλίνου. Την ασφάλεια, την ευμερία, την κοινωνική ανάπτυξη, τι απόψει του ε, παιδιού με βάση την ηλικία και την οριμότητά του. Αυτά υπάρχουν στο 6.3 συν η ταυτότητα του παιδιού, το κατά πόσο είναι ευάλωτο και οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να μεταφερθεί η διάρκεια διαμονής στο κράτος το οποίο βρίσκεται εκείνη τη στιγμή και οι άλλες χώρες στι οποίε έχει διαμείνει, η προσαρμογή του παιδιού στις ε, χώρες αυτές και η ανάγκη να αναπτυχθεί το παιδί. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη Και όταν έχουμε όλα τα στοιχεία ε, για το μείζον συμφέρον του παιδιού, τότε θα πρέπει να λάβουμε την απόφαση με βάση αυτό. Η αρμοστία επίσης πιστεύει ότι πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση από φορείς προστασίας του παιδιού που έχουν τη γνώση για να αξιολογήσουν τι είναι προς το συμφέρον του συγκεκριμένου παιδιού. Πιστεύουμε πρέπει να μην είναι το βασικό κριτήριο ε, για τον καθορισμό της ε, ευθύνης η, η φάση στην οποία βρίσκεται η αίτηση του παιδιού, ε, σε ποιο βαθμό έχει διεκπεριωθεί κτλ. Το βασικό σημείο αφετηρίας είναι ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει να μεταφερθούν εάν δεν είναι προς το συμφέρον τους. Στο παρελθόν ξέρουμε ότι είχαμε προβλήματα με καθυστερημένη πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, γιατί υπήρχε πρόβλημα με, την, το διορισμό του κηδεμόνα, υπήρχε πρόβλημα με την αμοιβαία αναγνώριση, υπήρχε πρόβλημα επομένως ε, με, το, με τη στέγη του, στέγαση του παιδιού και καμιά φορά το παιδί ήταν άστεχο μετά τη μεταφορά του για τις ε, δικονομικές ασφαλιστικές δικλείδες. Θα πρέπει το παιδί να του διοριστεί ένας κηδεμόνας στο συντομότερο δυνατό, ε, για να έχει τη δυνατότητα να έχει και προσωπική συνέντευξη που θα λάβει υπόψη το βαθμό οριμότητας, το ευάλωτο του παιδιού. Επίσης ε, ε, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που είναι ευαίσθητες με βάση τη διαδικασία. Και το βασικό είναι να μην, τα παιδιά τα οποία δεν έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου να μην, μπουν, να μην πέσουν ας πούμε, σε κάποιο νομικό λίμπο. Ευχαριστώ κυρία Κέσλε, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Προσφύγων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήμουν ένας από αυτούς που σώθηκε από το Σανσέρ. Ευχαριστώ λοιπόν για, την, για το καλωσόρισμα το ιδιαίτερο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα μιλήσω και εκ μέρους και άλλων χριστιανικών οργανώσεων που από κοινού χαιρέτησαν την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε τρία λεπτά δεν μπορούμε να καλύψουμε όλε τι πτυχέ του προβλήματο. Όσον αφορά τον κανονισμό του Δουβλίνου για τα συνόδευτα παιδιά, θα ήθελα να περιοριστώ σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε θερμά που για πρώτη φορά και για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εισηγήτρια για την έξοχη δουλειά τους είναι σπάνια ευκαιρία για μη κυβερνητική οργάνωση να ευχαριστεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά που έκανε. Και δράτω με τις ευκαιρίες να το κάνω αυτό, να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για όσα έκανε, διότι το κείμενο όταν θεσπιστεί τελικά και γίνει νόμος θα είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Έχω σύντομα σχόλια, διότι οι προλαλήσαντε ήδη κάλυψαν το θέμα. Η πρώτη Συμβούλιο για νέα παράγραφο 4β στο άρθρο 8 τη συμβάσεω του Δουβλίνου είναι μια νέα παράγραφο που θα λέει ότι εν είδη παρεκκλήσεως από την παράγραφο 4α το υπεύθυνο κράτος μέλος θα είναι εκείνο το οποίο ήδη έχει λάβει απόφαση καταρχήν σε πρώτη φάση όσον αφορά την ουσία κατά πόσο να αποδεχτεί η αίτηση για διεθνή προστασία εκτός αν δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού, του ανηλίκου. Έχουμε κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την πρόταση. Πρώτα απ' όλα, η νέα παράγραφος κατά κάποιο τρόπο ε, την απόφαση του δικαστηρίου την αντιστρέφει. Τη φέρνει τούμπα με άλλα λόγια. Σύμφωνα το δικαστήριο, μια επιστροφή Δουβλίνων γέννη δεν είναι προς το καλύτερο συμφέρον του παιδιού η πρόταση του Συμβουλίου θα το αντέστρεφε αυτό και θα έλεγε για συγκεκριμένη ομάδα συνόδευτων ανηλίκων η επιστροφή είναι εν γέννη προς το καλύτερον όφελος του παιδιού αν δεν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις συγκεκριμένη περίσταση. Άρα είναι το αντίστροφο, ακριβώς το αντίστροφο της αποφάσεως του, του δικαστηρίου. Δεύτερον, η παράγραφος ε, προβλέπει μακρύτερες και περιπλοκότερες διαδικασίες. Θα είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει κανείς σε κάθε περίπτωση κατά κάποιο, κάποιο άλλο κάτω μέλος έχει λάβει κάποια απόφαση επί της ουσίας ε, της αιτήσεως και όχι επί διαδικαστικού. Και θα ήταν δύσκολο ε, να διαπιστωθεί κατά πόσο η διαδικασία στον λόγο κράτος μέλος κάλυψε και καλύπτει τις ανάγκες του παιδιού και η επιστροφή στο κράτος μέλος να μην βλάπτει την αρχή που προστατεύει το καλύτερο συμφέρον του παιδιού. Θα υπάρξει αύξηση της γραφειοκρατίας, θα επηρεάσει τα παιδιά, τα οποία ήδη είναι πολύ ευάλωτα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι αυτό η πρόθεση του Ευρωπαίου νομοθέτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κέσλερ. Η κυρία Ζαβένσκα. Εκ μέρους της ΕΚΡΕ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω που καλέσατε την ΕΚΡΕ σε αυτή την ακρόαση σήμερα και να σας πω ότι χαίρομαι που εκπροσωπώ την ΕΚΡΕ, το Ευρωπαϊκό Νομικό Δίκτυο Ασύλου, που είναι ένα δίκτυο 500 δικηγόρων σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκπροσωπούνται από εμά. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα Έχουμε εκδώσει συγκριτικές εκθέσεις για το Δουβλίνο και έχουμε βοηθήσει και πολλούς δικηγόρους σε πολλά κράτη-μέλη ε, σε υποθέσεις που έχουν σχέση με το Δουβλίνο και την ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Υποστηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για το άρθρο 8 παράγραφος 4 και πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε εξαίρεση από την αρχή της μη μεταφοράς ε, που ε, προτείνουμε και εδώ και πολύ καιρό θα πρέπει να είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Η πρόταση της Επιτροπής είναι συμβατή με την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ενώ η πρόταση του Συμβουλίου μειώνει κάπως αυτή την, το εύρος αυτής της αρχής δεν καλύπτει το μείζον συμφέρον του παιδιού η πρόταση του Συμβουλίου κατά τη γνώμη μας και δεν λαμβάνει υπόψη την προστασία και την φροντίδα που απαιτούνται για τα παιδιά βάσει του άρθρου 24 ε, της Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα παιδιά και οι αιτούντες άσυλο, όπως και στη σχετική νομολογία, θα πρέπει να προστατεύονται και να προστατεύονται τα συμφέροντα των παιδιών. παρακολουθούμε την νομολογία μετά την απόφαση ΕΜΕΗ στα κράτη-μέλη και χαιρόμαστε διότι πολλά κράτη-μέλη αναγνωρίζουν αυτά τα σημαντικά θέματα. Ιδιαίτερα στα διοικητικά δικαστήρια, όταν αναφέρονται στην απόφαση MA, τονίζουν ότι κανένα παιδί δεν θα πρέπει να υπόκειται σε αλλαγή τοποθεσίας όταν μπορεί αυτό να αποφευχθεί. Στη διοικητική απόφαση 313 του Σάρλαντ αναφέρεται κάτι τέτοιο και επίσης θέλουμε να τονίσουμε ότι επειδή υπάρχει ο πολύ ευάλωτο χαρακτήρα των παιδιών, αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο κανόνα που προτείνεται από το Συμβούλιο μπορεί να δημιουργήσει περιτά εμπόδια για τα εμπλεκόμενα παιδιά. Ακόμη, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο να γίνεται αξιολόγηση του μείζωνος συμφέροντος του παιδιού και ειδικοί όροι θα πρέπει να ισχύουν Διαφορετικά θα μπορούσε να καταλήγει ε, αυτή η διαδικασία σε απάνθρωπη και υποτιμητική μεταχείριση για τα παιδιά. Ακόμη τονίζουμε ότι η αναδιατύπωση του κανονισμού του Δουβλίνου ήδη τονίζει την αρχή του μείζωνος συμφέροντος ε, των παιδιών όπως ήδη ανέφεραν οι συνάδελφοι. Ακόμη χρειάζονται διαδικαστικές εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους λόγω του ευάλωτου χαρακτήρα τους. Για να υλοποιηθούν αυτές οι εγγυήσεις υπάρχει υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται για να αξιολογείται το μείζον συμφέρον του παιδιού και αυτό θα πρέπει να είναι αντικείμενο παρακολούθησης και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζεβένσκα. Ο κύριος Μίτλικοφ, εκ μέρους της Επιτροπής Μάιζες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους της Επιτροπής Μάιερς, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε για να επαναλάβω τις απόψεις μας για το θέμα αυτό Είμαστε μια ομάδα ε, δικαστών, ε, δικηγόρων ε, στην Ολλανδία που έχουμε γνώση αυτών των υποθέσεων. Θα περιοριστώ σε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο αφορά την ανάγκη να εφαρμόσουμε πλήρως την απόφαση του δικαστηρίου. Μια, η απόφαση ή μάλλον η απόφαση, η πρόταση του, της Κομισιόν και η πρόταση του Συμβουλίου είναι ξεκάθαρη και υπάρχει εξαίρεση για ανηλίκους που ε, υποστηρίζει την ακαιρεότητα του συστήματος του Δουβλίνου ε, για να μειωθεί και ο κίνδυνος για το ανθρώπινο εμπόριο πρέπει να αποφασίσουμε να καταπολεμήσουμε το έγκλημα. Αυτό ακριβώς είναι το, ο στόχος του συστήματος. Νομίζουμε ότι κακώς θα θεωρούμε ότι οι διαδικασίες ασύλου είναι σωστές σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, πολλά κράτη-μέλη δεν μπορούν να εφαρμόσουν σωστές, ε, σωστά λειτουργούσε διαδικασίε όλοι οι αιτούντες άσυλο ε, που ταξιδεύουν σε αυτά τα κράτη-μέλη είναι θύματα. Και βέβαια οι ανήλικοι που είναι ακόμη πιο ευπαθείς ε, υποφέρουν περισσότερο. Ε, όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, η Επιτροπή μας σας ενθαρρύνει να αρνηθείτε να δεχτείτε οι ασυνόδευτοι ανηλικοί να παραμένουν εκτεθειμένοι και βάλλονται σε αυτά τα ανεπαρκή νομικά συστήματα. Και θέλω να υιοθετήσετε την έκθεση της κυρίας Βίξτρομ. Δεύτερον, την ανάγκη να τροποποιήσουμε το άρθρο 27 για την νομική προστασία για να σας δείξω την ανάγκη γι' αυτό, να σας δώσω ένα πραγματικό παράδειγμα ενός ανηλικού που ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του ε, διαμένει νόμιμα σε ένα άλλο κράτος μέλος, όμως ε, χρειάστηκε να... Ε, χρειάστηκε τόσος χρόνος για να επαληθευτεί αυτό που πέρασε η τριμήνη περίοδο και έτσι το παιδί δεν μπόρεσε να ξαναβρει τον πατέρα του. Ο κανονισμό αυτό δεν προβλέπει αντικά για αυτή την περίπτωση και έχω και άλλα τέτοιου τύπου παραδείγματα και δεν εξασφαλίζει ότι ε, διαφυλάσσεται το μείζον δικαστήριο, ε, δικαίωμα του παιδιού από το δικαστήριο. Το άρθρο 27 ε, θέλει να προβλέψει ένδικα μέσα και το, οι τροπολογίες 19 και 20 θα ευθυγραμμίσει τον κανονισμό με τη χάρτα. Επίσης, δεν θέλουμε να υπάρχει asylum shopping. Το άρθρο 25 της ε, διαδικασίας για τα ε, ένδικα μέσα ε, θα πρέπει να προβλέπει, προβλέπει μάλλον διαδικασίες ούτως ώστε να αποφευθεί το shopping του ασύλου. Υπάρχει νομική βάση για επιμερισμό των φακέλων και η μεταφορά περιορίζεται σε έξι μήνες και μέσα αυτούς τους έξι μήνες μπορείτε να ε, στείλετε φακέλους, ας πούμε, ε, από το ένα κράτος στο άλλο κράτος. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπουτεγέ από το Save the Children. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που καλέσατε το Save the Children να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις τροποποίησεις του κανονισμού του Δουβλίνου θα απηχήσω κάποιες εκφραστήσεις ανησυχίες, όμως είναι σημαντικό σημερινή συζήτηση να δούμε και ποια είναι η πραγματικότητα. Πέρα από τις νομικές διατάξεις σήμερα στην Ευρώπη, βλέπουμε αύξηση του αριθμού παιδιών που έρχονται στην Ευρώπη ετούντα άσυλο. Σύμφωνα με τις στατιστικές, να θυμηθούμε ότι έχουμε περίπου 26.000 παιδιά που έφτασαν στην Ευρώπη να ζητήσουν άσυλο. Μεταξύ αυτών 13.000 περίπου ασυνόδευτα παιδιά που έρχονται κυρίως από τη Συρία, την Ερυθρέα και άλλες χώρες που βρίσκονται σε φοβερή αναταραχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η συζήτηση να έχει το σωστό πλαίσιο σήμερα. Επιστρέφω στις τροποποίησεις. Θα εστιαστώ επί τριών πτυχών. Είναι σημαντικό να δούμε τη λογική που χρησιμοποιεί το Συμβούλιο ερμηνεύοντας την απόφαση του δικαστηρίου. Να δούμε και το κατά πόσο είναι εφικτό να εφαρμοστεί πρώτα Συμβουλίου και να συζητήσουμε και το θέμα της πρακτικής συνεργασίας. Τώρα, όσον αφορά τη νομική λογική που ακολουθεί το Συμβούλιο, θα πηχήσω εδώ τα όσα είπε το GRS που είπε ότι αντιστρέφεται η λογική της αποφάσεως του δικαστηρίου. Και θα ήθελα να τονίσω εκ νέου ότι η αφετηρία της λογικής του δικαστηρίου είναι η παραδοχή του, της άκρος ευάλωτης καταστάσεως των παιδιών που έτουν άσυλο. Και αυτή η, η άκρε, ε, το άκρον ευάλωτο της, της καταστάσεως τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο μέτρο του δυνατού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Συμβούλιο εξετάζει από ποιο στενή οπτική γωνία το ποιο είναι το μέγιστο συμφέρον του παιδιού και δεν λαμβάνει υπόψη και το χρόνο. Η αρμοστία για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ είπε ότι το μέγιστο συμφέρον του παιδιού είναι περιπλοκότατη έννοια και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες. Όπως πόσο καλά είναι το παιδί, κοινωνική του ανάπτυξη, η ασφάλειά του, οι απόψεις ε, των παιδιών ανάλογα με την ηλικία του, ηλικία της, οριμότητα και ποιο είναι το όλο ιστορικό και το περιβάλλον του παιδιού. Λοιπόν, πολλά έχουν υποθεί αλλά θα ήθελα να επιμείνω επί του σημείου που έθεσε συνάδελφος. Το τοπίο της προστασίας στην Ευρώπη δεν παρέχει αντίστοιχη προστασία παντού. Έχουμε κάτι μέλη που παρέχουν μεγαλύτερη προστασία και άλλες χώρε έχουν μεγάλα κενά. Το ότι ελήφθη μια απόφαση δεν είναι de facto αυτή καθεαυτή ένας παράγοντας που οδηγεί σε μεταφορά του παιδιού. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει συμφωνία όσον αφορά το, την κατάσταση κυδαιμονίας αλλά υπάρχει ένα σύστημα που περιπλέκει την όλη διαδικασία. Τέλος, υπάρχει ανάγκη η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διεθνή συνεργασία να παραμείνει. Βασικό αρχιτεκτονικό στοιχείο του Δουβλίνου. Οι μονάδες του Δουβλίνου σήμερα δεν είναι καλά εξοπλισμένες. Έχουν επιχειρησιακούς περιορισμούς. Άρα σημαντικότατο θα ήταν το τελικό κείμενο να διατηρήσει την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα θέλαμε το Κοινοβούλιο επιμείνει επί της ανάγκης εφαρμοστικών μέτρων ούτω ώστε να υπάρξουν διαδικασίες που θεσπιστούν πρότυπα και να καθορίζεται σαφώς και το πεδίο εφαρμογής και το πλαίσιο συνεργασίας. Ευχαριστώ κυρία Μακρέιαν. Και τώρα τελευταία παρέμβαση από τους ενδιαφερομένους η κυρία Άτκερα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, θα ήθελα και εγώ εν πολύ να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Μιλώ εκ μέρους ε, των ε, οργανώσεων του Ερυθρού Σταυρού. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πιστεύουμε ότι είναι μεταξύ των πιο ευάλωτων ομάδων και γι' αυτό έχουμε ειδικέ ε, υπηρεσίες για την φροντίδα αυτών των ασυνόδευτων ανηλίκων. Καλύπτουμε δραστηριότητες όπως ψυχοκοινωνική βοήθεια, περίθαλψη και στέγαση καθώς και ανθρωπιστική βοήθεια για να μπορέσουν να ζήσουν και να ενταχθούν ε, σωστά. Από την εμπειρία μας ε, είναι ιδιαίτερα έντονος ο ευάλωτος χαρακτήρας των συνόδευτων ανηλίκων και παρότι αυτό είναι γνωστό στα κράτη-μέλη, το επίπεδο ε, προστασίας και υποδοχής ποικίλει κατά πολύ στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάσαμε πολύ προσεκτικά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και χαιρετίζουμε την απόφαση του Δικαστηρίου και της Επιτροπής. Τονίζουν τον ευάλωτο χαρακτήρα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Συμφωνούμε ότι χρειάζεται μια ειδική προσέγγιση που προστατεύει τα παιδιά που είναι διαφορετική από τις αρχές που διέπουν το Ευρωπαϊκό Κοινό Σύστημα Ασύλου. Χαιρετίζουμε το ότι το σχέδιο έκθεσης του Κοινοβουλίου δείχνει ότι υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής. Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι να επικρατεί το μείζον συμφέρον του ανηλίκου σε κάθε περίπτωση. Να εξετάζεται συστηματικά λοιπόν και η διαδικασία για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους δεν θα πρέπει να παρατείνεται όταν αυτό είναι περιττό. Συμφωνούμε ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία ε, προστασίας, αλλά όταν υπάρχει ε, μεταφορά, ε, η μεταφορά θα πρέπει να εφαρμόζεται κατ' εξαίρεση. Ακόμη και όταν υπάρχει απόφαση σε άλλο κράτος πιστεύουμε ότι κατά κανόνα ο ανήλικος δεν θα πρέπει να μεταφέρεται εκτός εάν αυτό είναι προς το καλύτερο συμφέρον του ανηλίκου. Θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε εξαιρέσεις των κανόνα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες ε, του παιδιού και θα πρέπει το μείζον συμφέρον του ανηλίκου να είναι η κύρια να είναι το κύριο μέλημά μας και τονίζουμε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια. Πρώτον, η άποψη του ανηλίκου, ανάλογα με την ηλικία του και την οριμότητά του και αυτό είναι θεμελιώδες για να περιορίζεται ο κίνδυνος εμπορίου ανθρώπων. Θα πρέπει επίσης να φροντίζουμε τα θέματα επικινδυνότητας και να λαμβάνουμε υπόψη και τους παράγοντες επανένωσης των οικογενειών. Αυτό είναι θεμελιώδης για να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση. Θα ήθελα τέλος να τονίσω ένα σχετικό θέμα που είναι εξίσου σημαντικό, τη δυνατότητα κράτησης των ετούντων άσυλο και την εφαρμογή μεταφορών σύμφωνα με το σύστημα του Δουβλίνου. Πιστεύουμε ότι κατά κανόνα ποτέ δεν πρέπει να γίνεται κράτηση ανηλίκων. Θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι τωρινέ διατάξει σχετικά με την κράτηση, ώστε να είναι αναλογικές και να τηρούν ε, την, ε, να φροντίσουμε να γίνεται σεβαστή η ακαιρεότητα και η αξιοπρέπεια του ανηλίκου. Θέλουμε να ισχύσουν ε, τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ιδιαίτερα ε, και σε σχέση με την οδηγία για την υποδοχή. Επανέρχομαι τώρα στην σημερινή συζήτηση για το υπεύθυνο κράτος για την εφαρμογή ε, των μέτρων αυτών. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει κυρίως ε, να μην σκεφτόμαστε το ποιος πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη, αλλά το πώς θα πρέπει να έχουμε διαδικασίες φιλικές προς τα παιδιά που θα επιτρέπουν βιώσιμες λύσεις. Αυτό ώστε η προστασία των παιδιών να, και τα δικαιώματα των παιδιών να είναι στο επίκεντρο των μελημάτων μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, που ήρθατε στην Επιτροπή μας και μας είπατε αυτά τα σημαντικά στοιχεία. Θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές, καταρχάς στους κοιόδης εισηγητές και μετά στην εισηγήτρια. Κυρία Ματσόλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ομιλητές, τους καλεσμένους μας που θα να μιλήσουν. Η Σεσίλια είπε ότι επαναλαμβάνεται, αλλά θέλω να την ευχαριστήσω για τη δουλειά της, θέλω να την ευχαριστήσω για τις προσπάθειές της. Συντόνισε τις εργασίες με τους κοιόδης εισηγητές και θέλω να την υποστηρίξω μέχρι τέλους για όλες τις προσπάθειες που έκανε σε όλους τους ευρωπαϊκούς ε, στα ευρωπαϊκά νομοθετήματα, ειδικά σε, αυτή την, ε, σε αυτόν τον τομέα όπου προσπαθούμε να προωθήσουμε το συμφέρον του παιδιού. Όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, σήμερα μιλάμε για το τι μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε το μείζον συμφέρον του παιδιού. Ειδικά σε αυτό το τομέα, στο θέμα του ασύλου. Όπως είπε και η τελευταία ε, ομιλήτρια, και εγώ μιλάω για μια κατηγορία ανθρώπων που είναι πολύ ευάλωτη. Ξέρω ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης αυτή τη στιγμή είναι εν εξελίξει στη Μεσόγειο. Ακούμε πολλές ειδήσει, πολλά νέα. που μας, μιλάνε για αυτό το για αυτούς τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί, που είναι το αντικείμενο της σωστικής προσπάθειας. Η ομάδα μας δεν υπέβαλε τροπολογίες, ήθελα να σας πω, αλλά κάθε τροπολογία που υποβάλλεται στον κανονισμό μετά την απόφαση του δικαστηρίου ε, θέλω να πω ότι κάθε τροπολογία πρέπει να είναι ευσύνοπτη, ξεκάθαρη, ούτως ώστε να χύνει περισσότερη ενάργεια έτσι, στο θέμα αυτό. Πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των παιδιών. Ευχαριστώ. Ρομπέρτα. Η κυρία Σίμπελτ. Θα εκπροσωπήσει την κυρία Γκυγιόμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ομιλώ εξ ονόματος της δυσηγήτριας Σιβή Γκυγιόμ που δυστυχώς δεν είναι παρούσα σήμερα. Όπως κυρία Μετσόλα, και η κυρία με ευχαριστεί την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε και την επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων πάντα ήταν και είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, πολύ λεπτό θέμα. Από τη μία έχετε εκείνους που επιμένουν ότι είναι πολύ ευάλωτα τα παιδιά και ότι πρέπει να προωθήσουμε τις ασφαλιστικές δικλίδες που απαιτούνται για να τα προστατεύσουμε. Και από την άλλη Έχουμε εκείνους που κατ' επανάληψη φοβούνται από την πιθανότητα εισβολής ε, τέτοιων ανηλίκων στην Ευρώπη, αν έχουμε τέτοια μέτρα. Όπως υπόθηκε πολλές φορές, υποστηρίζω, υποστήριξη μάλλον της πρότασης της Κομισιόν ε, είναι ε, γιατί είναι καθαρή απεικόνηση της ε, άποψης που έχει το δικαστήριο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τη λογική που υπάρχουν ε, και την ε, γενική οικονομία του κειμένου. Ω και συγγήτρια, αποφάσισα λοιπόν ακριβώ γι' αυτό να μην υποβάλω καμία τροπολογία, ούτω ώστε να φτάσουμε σε μια ευρωπαϊκή θέση που να είναι ο πιο κοντά στην πρόταση τη Κομισιόν και κατά συνέπεια και στην απόφαση του δικαστηρίου. Η νομική διευκρίνηση είναι ακόμα περισσότερο αναγκαία όταν βλέπετε πόσο πολύ η αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές ερμηνείες στα πλαίσια του κανονισμού του Δουβλίνου. Πέρα από την νομική διευκρίνηση, το ευάλωτο των παιδιών, εδώ λαμβάνεται πλήρως υπόψη και έτσι θα αποφύγουμε περιτές και επιζήμιες μεταφορές ανηλίκων από το ένα κράτος στο άλλο. Αυτά από την σκιώδη συγκητριά μου. Και επιτρέψτε μου και μένα μία πρόταση σε απάντηση αυτά που ακούσαμε από το Συμβούλιο. Θέλετε μία γρήγορη απόφαση. Είναι πιθανό. Πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα επιτέλους ότι οι Ευρωπαίοι δεχόμαστε τους ανθρώπους που φεύγουν από τον πόλεμο και από άλλες ε, καταστροφές τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες που χρειάζονται. Φτάστε λοιπόν στο επίπεδο της θέσης ε, της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου και τότε θα έχετε τη γρήγορη απόφασή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του σκιώδου συζητητού μας του Κίρκοπ ευχαριστώ την κυρία Βίκστρομ. Το μέγιστο συμφέρον του παιδιού πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη, εξυπακούεται αυτό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην δημιουργήσουμε τέτοια νομοθεσία και διαδικασίες που να ενθαρρύνουν ε, την επιδίωξη καλύτερου μέρους για ε, άσυλο και να μεταφέρονται οι άσυλο από μια χώρα σε άλλο κράτος και άλλα τέτοια ανεπιθύμητα φαινόμενα. Θέλουμε το συμφέρον του ανηλίκου να προστατεύεται, είναι και θέμα αξιοπιστίας και νομιμότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών περιασύλου. Η... Μία αναγκαία μεταφορά παιδιών μεταξύ κρατών μελών πρέπει να αποφεύγεται. Πρέπει όμως να υπάρχει δυνατότητα να επιστρέφει ένας ανήλικος στο κράτος μέλος εκείνο το οποίο υπέβαλε την πρώτη αίτηση. Αν εκείνο το κράτος μέλος έχει ήδη αξιολογήσει κατ' ουσίαν κατά πόσο ο ετών ή ετούσα ε, δικαιούται διεθνούς προστασίας. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος ότι κάποιο άτομο μετακινείται ή μεταφέρεται ελαθρέα σε άλλο κάτω μέλος, εκείνο όπου τα κριτήρια για τη χορήγηση προστασίας ή κανόνες περί οικογενειακής επανένωσης είναι πλέον ευνοϊκοί. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ένα κάτω μέλος όπου είναι παρόν ο ετών θα είναι σε καλύτερη θέση να αξιολογήσει επακριβώς και ταχαίως ε, τα επιχειρήματα της δεύτερης αιτήσεως εν συγκρίση με το κράτος μέλος εκείνο που εξέτασε την πρώτη αίτηση. Συμφωνώ με τον κύριο Νίτλκοπ και άλλους. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Οι διαδικασίες και τα πρότυπα υποδοχής που ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Δεν έπρεπε να γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν προβλέπει κάτι τέτοιο ο κανονισμό του Δουβλίνου. Πρέπει να είναι εξομοιωμένα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρξει κάποιος έλεγχος ε, και να δουν ποιο είναι υπεύθυνο για αυτές τις διαδικαστικέ ελλείψεις και διαφορές. Ευχαριστώ κυρία Μπιόρκ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς πρέπει να πω ότι ε, πολλά μπορούμε να πούμε για το Δουβλίνο και ελάχιστα θετικά. Υπάρχουν ε, πολλές παράλογες πτυχές που περιέχονται. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε επί των νομοθετικών τροποποίησεων που έχουμε μπροστά μας. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βίκστρομ που εργάστηκε άοκνα. Ε, σε επαφή με όλους. Εξετάσαμε με εκδητικό φακό τις λεπτομέρειες. Πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει να παραμείνουμε όσο πιο κοντά γίνεται στην απόφαση του δικαστηρίου με κάποιες αλλαγές, ε, τροπολογίες που θα κατατεθούν, θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα όπου μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για τα παιδιά που ετούν άσυλο. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προσπάθειες που έκανε και που μας βοήθησε να συμφωνήσουμε και θα προχωρήσουμε σε προσπάθειες να καταλήξουμε σε ενεντικές ε, τροπολογίες. Είναι ένα πρώτο βήμα, σημαντικό βήμα όμως αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προβλέψουμε ένα καθεστώς εξαιρέσεων για τα παιδιά. Και θέτω το ερώτημα, ποιος είναι ο αριθμός αυτών. 26.000 παιδιά, ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά που έρχονται. Ε, είμαστε απογοητευμένοι από τις συζητήσεις στο Συμβούλιο δεν θα πρέπει να απομακρυνόμαστε από την απόφαση του δικαστηρίου. Είχαμε συμφωνία το 2013 και πρέπει να γίνει σεβαστή συμφωνία. Η συγγήτρια το σέβεται αυτό και οι σκιώδεις συγγητές θα σεβαστούμε αυτή την απόφαση. Δεν δεχόμαστε τη στάση του Συμβουλίου που πηγαίνει αντίθετα στις ε, απόψεις των προσκεκλημένων των εμπειρογνωμόνων. Έχουμε εμπειρογνώμονες εδώ και άλλους, που, αυτούς που μίλησαν και άλλους που μας γνωστοποιούν τις θέσεις τους. Δεν θα πρέπει να κινούμεθα κατά της αποφάσεως του ΔΕΚ, ούτε κατά της συμβάσεως του ΙΕ για την προστασία των ανηλίκων. Ε, θα ντροπή, ντροπή στο Συμβούλιο. Πρέπει να επιστρέψετε στο, στις διαπραγματεύσεις και να δείτε ποια είναι η θέση σας. Δεν, δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών. Θα πρέπει να βλέπουμε ποιο είναι το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών. Και θα συνεργαστούμε με την εισηγήτρια θα παραμείνουμε όμως στεναροί στις πεπιθήσεις μας. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς και να υπονομεύουμε τα συμφέροντα 26.000 παιδιών που έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πραγματικότητα και η κατάσταση αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά. Εκτίθενται στο χείριστο, στις χείριστες συνθήκες αυτά τα παιδιά. Ό,τι χειρότερο που θα μπορούσε να του συμβεί. Λοιπόν, θα πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στις θέσεις μας και να τα προστατεύσουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Λαμπέρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να προσθέσω τη φωνή μου στους προλαλήσαντες που ευχαρίστησαν την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει και σας ευχαριστούμε και για ε, ε, τους εμπειρογνώμονες που προσκαλέσατε και ακούσαμε σήμερα. Το Δουβλίνο 2 ήταν ασαφές όσον αφορά τις ευθύνες για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Στην προηγούμενη θητεία υπήρξε μια, συμβουλή, μια συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι θα δεχόμασταν την απόφαση του δικαστηρίου για να έχουμε κάποια σαφήνεια. Τώρα έχουμε αυτή τη σαφήνεια και όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, θεωρώ απογοητευτικό το ότι το Συμβούλιο συνεχίζει να θέλει να συζητά το θέμα αφού έχουμε εξαντλήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Όπως ακούσαμε από την Επιτροπή Μάιζερ σήμερα και όπως γνωρίζουμε και όπως το αναγνωρίζει και ο κανονισμός, υπάρχουν ε, διαφορετικά στοιχεία στο πώς ε, εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη το κοινό σύστημα ασύλου. Το γνωρίζουμε όλοι. Ήταν μεγάλη συζήτηση που είχαμε κάνει στην προηγούμενη θητεία για την υλοποίηση του κανονισμού του Δουβλίνου και επομένως και αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Η ομάδα μου δεν υπέβαλε τροπολογίες στην έκθεση αυτή, διότι θέλουμε να υπάρχει ως το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια και συνένεση για την θέση του Κοινοβουλίου, ούτω ώστε να μην υπάρξει στη συζήτησή μας με το Συμβούλιο καμία έλλειψη σαφήνειας. Συμφωνώ απολύτως με την κυρία Σίπελ που μας είπε ότι αν το Συμβούλιο θέλει να αλλάξει κάποια απόφαση, ε, αν, θέλουμε μια γρήγορη απόφαση, το Συμβούλιο μπορεί να λάβει μια σύντομη απόφαση, ούτως ώστε να μην εκτίθεται τα παιδιά σε αυτή την κατάσταση με όλους τους κινδύνους που τη συνοδεύουν. Ας κλείσουμε λοιπόν το θέμα των συντομών Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Λάμπερτ. Άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν το λόγο. Κυρία Βίνμπεργ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις ε, πληροφορίες. Έχω καταθέσει μια τροπολογία που λέει ότι όταν τα παιδιά, οι νέοι, γιατί μερικές φορές δεν είναι παιδιά, αλλά νέοι, υποβάλλουν πολλές αιτήσει σε πολλά κράτη-μέλη. Αυτό είναι, πάρα, είναι περιττό για τις μεταφορές. Ε, σκέφτομαι ότι υπάρχουν οι διακινητές οι οποίοι μεταφέρουν παιδιά από κράτος σε κράτος. Και έτσι συσσωρεύονται σε κάποια κράτη παιδιά. Το βασικό είναι ότι πρέπει να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τα παιδιά. Αλλά στη Σουηδία, Φερρυπίν, βλέπουμε ότι Έχουμε μόνιμες άδειε που δίδονται σε Σύριους. Έχουμε 7.000 νέους ασυνόδευτους και, πήραμε και δεχτήκαμε και 7.000 ε, πέρυσι. Δεν θα πρέπει να γίνουμε φυτόριο για τους ε, διακινητές, δηλαδή όπου οι διακινητές θα έρχονται και θα συσσωρεύουν παιδιά, θα ξεφορτώνουν παιδιά. Ευχαριστώ. Κανένας άλλος συνάδελφος δεν θέλει να παρέμβει, άρα η Σεσίλια. Ευχαριστώ. Απευθύνομαι στους ε, καλεσμένους μας. Τους ευχαριστώ για τις πολύτιμες συνεισφορές τους που θέτουν ε, σημαντικά θέματα για το βέλτιστο συμφέρον και την προστασία των ανηλίκων που όλοι πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν ε, εξετάζουμε αυτό το κείμενο που έχουμε μπροστά μας. Στρέφομαι προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν και προς τους κοιόδες εισηγητέ και τους ευχαριστώ όλους για τις προσπάθειές τους επί του φάκελου αυτού και για όλες τις α, που άκουσα. Ε, καλωσορίσω τις τροπολογίες των συναδέλφων. Είναι προς την ίδια κατεύθυνση με το πνεύμα του, του κειμένου μου θα συζητηθούν στη συνάντηση των σκιωδών. Ε, θα σας στείλω email όταν ε, αποφασίσουμε την ημερομηνία. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, αλλά σύντομα θα σας ενημερώσω. Θέλω να επανέλθω σε ένα θέμα τώρα που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι μεταφορές γενικά είναι χρονοβόρες και δεν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Δεν τους χτίζει ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί το παιδί πρέπει να κάνει νέε προσπάθειε για να ξαναχτίσει τη ζωή του. Στην ε, οδηγία για τι συνθήκε υποδοχή έχουμε αναφέρει ότι οι αλλαγέ τη κατοικία των ασυνόδευτων ανηλίκων θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο αναγκαίο. Η νέα οδηγία για τα διαδικαστικά μέτρα μιλά ε, για την ε, διεκπαιρέωση των αιτήσεων μέσα σε έξι μήνες ασύλου δηλαδή. Ε, όμως η μεταφορά χρειάζεται συχνά περισσότερο χρόνο από έξι μήνες. Επομένω οι ασυνόδευτοι ε, θα έχουν πρόσβαση σε μια πιο γρήγορη διαδικασία εάν εξεταστεί η αίτησή τους στο κράτος μέλο που είναι παρόντα. Ε, βέβαια υπάρχει το αντεπιχείρημα ότι αν υπάρχει πρωτόβαθμη απόφαση σε ένα άλλο κράτος εκεί θα πρέπει να εξεταστεί. Ε, όμως ε, εκεί που είναι ανοιχτή η υπόθεση του, του ανηλίκου, ε, θα πρέπει εκεί να επιστραφεί ο ανήλικος. Ε, και επομένως, το πρόβλημα είναι ότι επειδή η διεκπαιρέωση της υπόθεσης του φακέλου παίρνει περισσότερο χρόνο από τους έξι μήνες, είναι πολύ δύσκολο. Και το θέμα είναι, εάν ανοίξει μια νέα ε, υπόθεση ε, στο κράτος μέρος είναι παρόν το παιδί, ε, μπορεί η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη. Υπάρχει κίνδυνος ότι το δικαστήριο θα θεωρήσει ότι αυτή η διάταξη είναι παραβίαση της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα έχουμε ε, πολλές ε, υποθέσεις στο δικαστήριο. Για να αποφύγουμε τις ε, καταχρήσεις, το δικαστήριο και η νομοθεσία έχουν βρει μια λύση. Αν μια αίτηση στο δεύτερο κράτος είναι ίδια με την αίτηση που έχει υποβληθεί ε, στο πρώτο κρατός μέλο που έχει κλείσει η διαδικασία, το δεύτερο κρατός μπορεί να θεωρήσει ότι η αίτηση είναι μη παραδεκτή. Θα πρέπει να δώσει νέα στοιχεία στο, στη νέα αίτηση ο φάκελο θα πρέπει ίσως να μεταφερθεί από το πρώτο στο δεύτερο κρατοσμέλος και ενδεχομένω, τα βασικά στοιχεία θα πρέπει επίση να μεταφραστούν. Αν συγκρίνουμε με τη μεταφορά του ανηλίκου στο πρώτο κρατοσμέλος, αυτό θα οδηγήσει σε μια διοικητική διαδικασία που θα χρειαστεί κάποιο χρόνο. Σίγουρα. Όμως, ο ασυνόδευτος ανήλικος θα έχει τουλάχιστον ε, τη δυνατότητα να αποφύγει την περαιτέρω μεταφορά και όλες τις αφεβαιότητες που συνοδεύουν αυτή τη μεταφορά. Και μια μακρά περίοδο χωρίς μέλλον και χωρίς προοπτική. Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους με βάση τον κανονισμό του Δουβλίνου. Μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση της έτασης για τη διεθνή προστασία. Αυτή η συνεργασία συνάδει επίσης με το άρθρο 4 της Συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαστήριο έχει εξετάσει το συμφέρον του ασνόδευτου ανηλίκου και θεωρεί ότι είναι σημαντικότερο από το πιθανό βάρος για την επανεξέταση μιας άλλης αίτησης από ένα άλλο κρατός μέλος. Αντί λοιπόν να θεωρούμε τους ανήλικους ότι είναι στο ίδιο επίπεδο με τους ε, ενήλικους αιτούντες, το δικαστήριο είπε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες του κεκτημένου ασύλου για να εξετάζουν τις ίδιες αιτήσει. Ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί ίσως δεν το είπα ευκρινώς την πρώτη μου παρέμβαση. Αλλά αυτή είναι η άποψη που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Τονίζω ακόμα μια φορά ότι σας ευχαριστώ για τις συνεισφορές σας και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπούμε σε λεπτομέρειες παρατηρήσεις, αλλά μπορούμε και τώρα και αργότερα να συζητήσουμε με τους σκιώδεις συγητές, αλλά και με άλλους συναδέλφους που μπορεί να ενδιαφέρονται από αυτό το πολύ σημαντικό αλλά πολύ λεπτό θέμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Σεσίλια. Ευχαριστώ για τη δουλειά που έκανες. Και τώρα, τα τελευταία δύο σημεία της ημερήσιας διάταξής μας για την απογευματινή συνεδρίαση έχουν αναβληθεί. Άρα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας και να σας το ανακοινώνω αυτό διότι το πρώτο σήμα της ημερήσιας διάταξης αναβάλλεται επίσης για αύριο το πρωί. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει λοιπόν στις 10 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ λοιπόν και θα τα ξαναπούμε στις 10 το πρωί αύριο. Γεια σας.